Υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις σας και η Πρόεδρος αλλά και η συγγήτρια της ομάδας Ε, η κυρία Στρίφλερ είχε μια υποχρέωση, συμμετέχει ως παρατηρήτρια σε κάποιες εκλογές αλλά ανταυτής θα μας προσφέρει τα συμπεράσματα ο κύριος Μπέρμαν. Έχετε το λόγο κύριε Μπέρμαν. Η ομάδα εργασία ε, θέλω να σα πω ότι στις 23 Δευτέρου συζήτησε αυτή την τέταρτη δέσμη μέτρων από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια τη ε, Διατροφική ε, ασφάλεια σε Ζάμπια, Κόγκο και άλλες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το υπήρξε πνεύμα συνεργασία και πρέπει να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενημέρωσή τη. Όμως, επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ομάδα εργασία ε, μπορεί να αποφανθεί μόνο επί τη βάση των εγγράφων που υποβλήθηκαν δυνάμει της επιτροπολογίας και άλλα γιατί δυστυχώς λείπανε κάποια πάρα πολύ βασικά στοιχεία. Επομένως δεν είχαμε πλήρη ενημέρωση όσον αφορά το τι θα πρέπει να κάνουμε. Οπότε και εμείς τώρα θα πρέπει να παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια επιτροπολογίας να μας υποβάλει όλη την σχετική τεκμηρίωση. Τανζανία, Τόγκο, ε, Κομόρος. Ε, συνεχίστηκε η γραμμή πλεύσης του Νοεμβρίου για την τρίτη δεσμή μέτρων, τόσο ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτές τις προτάσεις με τα μέτρα που, για την πολιτική που έχουμε όσον αφορά τη διατροφική επάρκεια και επίσης θεωρούμε ότι η τεκμηρίωση δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει αιτιώδη σχέση μεταξύ των, των δεδομένων και των, ε, των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη δημοσιονομική πτυχή και θα πρέπει να δούμε πώς το πρόγραμμα θα καλύψει και την ε, ε και αυτό θα πρέπει να αναλυθεί καλύτερα στο δελτίο ανάληψης δράσης. Επομένω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σα ασφαλίσουμε το, το πώ θα ανταποκρίνεται αυτό το πρόγραμμα στου στόχου τη διατροφική επάρκεια. Παρά το όσο μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί οι διαπραγματεύσει με τι κομμόρε συνεχίζονται, θεωρεί η ομάδα εργασία ότι έχουμε κάτι πια πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, όπω το κριτήριο τη εποπτεία για την εκταμή χρημάτων. Θα πρέπει όλα αυτά να διατυπώνονται στην, ε, στο, στο, στο δελτίο ανάληψη δράση και θεωρούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει τόση ασαφή τόσο ώστε δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε το πώς θα ενταχθεί αυτό το πρόγραμμα στους ε, στόχου του συγκεκριμένου και πώ θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα μέτρα τα οποία ε, χρειάζονται για να υπάρχει διατροφική επάρκεια. Επομένω, ε, έχουμε κάποια συμπεράσματα που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο κειμένου το οποίο να καλύπτει τα βασικά σημεία τα οποία έχουν αναλυθεί και ζητούμε επίση στο σχέδιό, στο ναι, θα πρέπει να αναθεωρήσει το, το, το, το, το δελτίο η Επιτροπή ούτως ώστε να μπορέσει να καλύπτει περισσότερο την αναγκαιότητα της, ε, διατροφικής, της των μέτρων για διατροφική ασφάλεια Με δεδομένα αυτά λοιπόν τα οποία διατυπώνουμε στην, ε, στο, στο σχέδιο κειμένου μας, περιμένουμε στα πλαίσια της Επιτροπολογίας να υποβάλει αυτά τα οποία ζητούμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω όπω έχουν τα πράγματα, καλώ του συναδέλφου να εγκρίνουν αυτό το σχέδιο ψηφίσματο το οποίο εκπώνησε η ομάδα εργασία, αυτό το οποίο σα έχει υποβληθεί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμεί ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρο και τώρα το λόγο έχουν τα μέλη τη Επιτροπή μα. Έχει κάποιε παρατηρήσει. Μπέρμαν. Ως μέλος θα ήθελα να προσθέσω ότι νομίζω ότι δεν μιλούμε για τροφική διευκόλυνση, ασφάλεια. Το πιο σωστό είναι να δούμε πώς τα κονδύλια που προβλέπονται για αυτό το στόχο, πώς θα αξιοποιούνται για κάποιο σκοπό που δεν θα είναι ασαφής. Δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο η πρόεδρος. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε και εσάς κύριε Μπέρμαν για τα καλά σας λόγια όσον αφορά το πνεύμα συνεργασίας με εμάς όταν συναντηθήκαμε με την ομάδα εργασίας θα πρέπει να σας πω για τη διαδικασία δύο λόγια και οι συνάδελφοι που παρίστανται να σας συμπληρώσουν τυχόν λεπτομέρειες. Βεβαίω και θέλουμε να σας καλύψουμε με αυτό που σας απασχολούν και όταν ε, παρουσιάσουμε την πρότασή μα, προσπαθήσαμε όσο ήταν ε, δυνατόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση ούτως ώστε να έχουμε μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων. να ακούσουμε τις απόψεις σα τα σχόλιά σα. και να λύσουμε τα τυχόν προβλήματα σε ένα τέτοιο ε, πνεύμα φιλικό και συνεργασίας. Επίσης, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να έχουμε μια γρήγορη ανταλλαγή απόψεων να σας ενημερώσουμε τυχαίως γιατί από ό,τι καταλαβαίνω επί τη βάση των όσων συζητήθηκαν την τρίτη περσμένη εβδομάδα έχουμε όλες αυτές τις παρατηρήσεις που σας διαβάσαμε την Παρασκευή το πρωί. Ετσι θεωρείτε ότι δεν αρκούν αυτά τα οποία εμεί υποβάλαμε, οπότε και εμείς ε, θα δούμε πώ είναι δυνατόν να έχουμε ε, μια πιο στενή ανταλλαγή όπω πώς να αξιοποιήσουμε τους τη επικοινωνία και ελπίζουμε ότι η αντιδράση μας πιο γρήγορα. Έτσι ήλπισα εγώ. Και είχαμε μέχρι τις 23 Μαρτίου ούτως ώστε να επιλύσουμε τις τυχόν διαφορές. Αν είχατε κάποια πρόταση επίση πριν τις 23 Μαρτίου Οπότε θα μπορούσε να υπάρχει μια, μια επιστολή σχετική με το τι σας προβληματίζει. Εξετάζουμε τώρα τις ε, τροπολογίες για το δελτίο δράσης και Τώρα θα δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο εξ αριστερών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ομάδα εργασίας που μας δίνεται αυτήν την δυνατότητα να σας πούμε τι έγινε στη συνέχεια της τρίτης δέσμης το Νοέμβριο. Προσπαθήσαμε να σας καλύψουμε και γι' αυτό και κάνουμε κάποιες βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά τη συμφωνία με το Μαλάουι. Επί τη βάση των δικών σας παρατηρήσεων προσπαθήσαμε επίσης να κινητοποιήσουμε και το γραφείο μας εκεί, ούτως ώστε έγκαιρα να κάνουμε αυτό το οποίο ζητήσατε. Ε, όντως θα πρέπει το δελτίο να βελτιωθεί και αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι θα πρέπει να ακολουθείται ταχεία διαδικασία για τέτοια θέματα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας τόσο ώστε να επιφέρουμε τις αλλαγές που θέλετε στο δελτίο δράσης. Μπέρμαν. Α, για τις κόμμαρες. Λίγα εκατομμύρια ευρώ είναι. Δεν είναι τίποτα τρομερό το οποίο διακυβεύεται, αλλά για πέστε μου, τι σας έκανε να χρησιμοποιήσετε υποτύπων γενική δημοσιονομική βοήθεια στα χρήματα που θα αφορούσαν τα είδη διατροφής δεν καταλαβαίνω πώς αυτό το οποίο προτείνεται σχετίζεται με την προσπάθεια εξασφάλισης διατροφικής επάρκειας. Όπως είπαμε τον Νοέμβριο και το επαναλάβαμε την προηγουμένη εβδομάδα η γενική δημοσιονομική υποστήριξη είναι κάτι που το προωθείτε και εσείς εδώ από το Κοινοβούλιο γιατί είπαμε ότι θα πρέπει οι επιλέξιμες χώρες να υποστηριχτούν και οι Κομορές είναι μια τέτοια περίπτωση επομένω. αυτή η υποστήριξη είναι ένα μέσον βοηθείας ούτως ώστε να αντισταθμίσουμε αυτά τα οποία έχουν δαπανηθεί λόγω της ανόδου των τιμών. Και τώρα θέλουμε πώς θα έχουμε κάποιους δείκτες επιδόσεων Αυτά συζητούμε με την κυβέρνηση για κάποιες δαπάνες οι οποίες έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό. Οπότε αφού τα συζητήσουμε θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διασκεδάσουμε τις αμφιβολίες σας. Βεβαίω, αν υπάρχει περιθώριο λιγμών θα σας ενημερώσουμε. Ο επόμενος. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. ασχολούν με θέματα ανάπτυξης και θα ήθελα να προσθέσω στα όσα είπαν ε, οι συνέλφοι από την άλλη Γενική Διεύθυνση. Σας είπαμε ήδη στα έγγραφα που διαβάζουμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε για ομικά τις κομμόρες και ο λόγος είναι ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε αυτό το οποίο χρειάζεται μια που δεν υπήρχαν και πάρα πολλά χρήματα διαθέσιμα και οι εναλλακτικέ θα ήταν να δούμε μήπως μπορούν οι διεθνείς φορείς να δώσουν κάτι για ότι αυτό είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε ε, τα κονδύλια που έχουμε για αυτήν τη χώρα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρος, γνωρίζουμε ότι ε, πιέζει ο χρόνος πάρα πολύ σε τις διαδικασίες, οπότε θα πρέπει σήμερα να γίνει η έγκριση του κειμένου και να υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Υπάρχει σχέση ψηφίσματος, να το προσθέσει ο κύριος ε, Μπερμάν και κατόπιν να γίνει η ψήφιση. Nous avons nous avons entendu qu'il y avait des difficultés détectées par notre Όμως, μας ε, είπε ο κ. Μπερμάνο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και δεν ξέρω τώρα συμφωνείτε να προχωρήσουμε. Κύριε Μπέρμαν, λυπάμαι πρόεδρε, αλλά δεν με έχει πείσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι το θέμα είναι τόσο σοβαρό τόσο δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε τόσο επιφανειακά. Δεν με έπεισαν με την απάντησή τους. Τι θα γίνει, θα περιμένουν, δεν θα έρθει ποτέ αυτή η βοήθεια. Τι θα γίνει με την γεωργική παραγωγή. Πρόεδρος. Τι θα κάνουμε. Προχωρήσουμε σήμερα με τόσο πρώτη ομάδα εργασία και να δούμε κατά πόσο θα, θα μπορέσουμε να έχουμε για αυτή τη διατροφική διευκόλυνση, την δημοσιονομική στήριξη. Α, καλά. Τότε εγκρίνεται. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ, να σηκώσουν το χέρι. Monsieur vous souhaitez la parole Κύριε Γκέρνς, θέλετε το λόγο. Νομίζω ότι ήθελε να πει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τόσους υπαλλήλους εδώ. Μπορούμε να ακούσουμε και άλλες ε, επεξηγήσεις. Ναι, βέβαια, εγώ νομίζω ότι τέλειωσε η Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος να περιμένουμε και άλλα έγγραφα, γιατί ε, έχουμε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς. Κομισιόν, έχετε κάτι να πείτε που δεν είπατε, κάτι, κάτι νέο σε σχέση με αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Γιατί βλέπετε ότι τώρα διακόψαμε τη δικασία της ψήφισης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Προείπα ότι θέλουμε να προχωρούμε επί τη βάση διαλόγου μόνο. Και θεωρούμε ότι το Κοινοβούλιο επιμένει ότι επιδέχεται βελτίωση η κατάσταση και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε να συμμορφωθούμε αυτό το οποίο ζητείτε. Και σας τονίζω ότι η διαδικασία η οποία προβλέπεται λέει ότι θα πρέπει κάτι το οποίο προτείνουμε να καλύπτει όλα τα μέτρα. Και αυτή η τέταρτη δέσμη είναι ευρύτερη από αυτό που ζητούν οι κομμόρες. Και δεν θέλουμε να μπλοκαριστεί όλο το πρόγραμμα επειδή υπάρχει μια επιμέρους διαφωνία. άλλα. Άρα αυτό το δελτίο που σας προβληματίζει ε, να το καλύψουμε αλλού και να χρησιμοποιήσουμε τις, τα αντίστοιχα κονδύλια για άλλο σκοπό. Πάντως, σας ε, ακούμε και θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Και καταλαβαίνουμε ότι ο κ. Μπέρμαν δεν έχει καλυφθεί με αυτά τα οποία άκουσε. Γέλνες. Επομένως, μετά αυτές τις χρήσιμες επεξηγήσεις θα βγάλουμε τις κομόρες και τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε στο κείμενο. Και εγώ συμφωνώ με αυτήν την λύση. Υπάρχει όμως συγκεκριμένη προθεσμία, λέει ο κύριος Μπέρμαν. Καταληκτική ημερομηνία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται να γίνει αυτό, τότε και εμείς μπορούμε να επεξεργαστούμε την περίπτωση που αφορά τις κομμόρες και να μην μπλοκάρουμε τις άλλες χώρες για να κινηθούμε και μέσα στα πλαίσια μας. Ναι, επιβάλλεται να τηρήσουμε αυτή την προθεσμία. Επομένω, θα ψηφίσουμε τώρα το κείμενο. Και αφήσουμε το δελτίο για τις κομμόρες εκτός συγκέρδυνση. Αν αποφασίσουμε σήμερα θα Έχουμε επομένω τι, την πρόταση Κομισιόν πλην κομμόρε. Ωραία. Να ψηφίσουμε από αυτού. Πρόταση Κομισιόν πλην κομμόρε. Και το θέμα το συζητήσουμε περαιτέρω, τόσο να καλύψουμε όλους όσοι έχουν κάποιε σκιέ εμβολίας. Αυτό θα πρέπει να γίνει αν θέλουμε να έχουμε ψηφίσμα. Μπέρμαν. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε αφού έχουμε αφαιρέσει τις κόμμορες. Αναφέρεται τουλάχιστον πέντε φορές Άρα θα πρέπει καλύτερα να ξαναδούμε μετά τη συνεδρίαση. Και αύριο οι συντονιστές να αποφασίσουν. Δεν ξέρω αν γίνεται. Δεν θέλω να αποφασίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Mm. Πρόεδρος, εάν όμως δεν αποφασίσουμε σήμερα η μόνη λύση είναι να έχουμε στο Στρασβούργο μια έκτακτη συνεδρίαση. Σαν Όμως, δεν καταλαβαίνω. Μέσα στην ψηφοφορία έχουμε προφορική τροπολογία της ε, Κομισιόν. Να συνεχίσουμε την, την ψηφοφορία. Και αν θέλουμε να γίνει μια τροποποίηση του κειμένου πριν την ε, ολομελία αλλά, αλλά αυτό δεν είναι σωστή διαδικασία. Το να βγάζουμε ένα κείμενο, να έχουμε προηγή τροποποίηση κομισιών, μια που έχει γίνει κάποια διαδικασία. Πρόεδρος. Τότε, να ψηφίσουμε το κείμενο ακριβώ ω έχει. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι s'abstient. Αποχές. Εγκρίνεται το κείμενο. Τώρα το 13. Voilà. Nous allons aborder maintenant le point 11 de notre ordre. Πάμε τώρα στο 11. Κλινικές δοκιμές σε αντισόμενες χώρες. Ακούσουμε κάποιου εμπειρογνώμονε. Πέρσι είχε γίνει από την Επιτροπή μα μια τέτοια μελέτη και καταλήξαμε σε κάποια ανταλλαγή απόψεων. Και έχουμε τώρα κάποιε συστάσει κατά αυτή τη ε, μελέτη και στη συνέχεια αυτών τώρα θα τα συζητήσουμε. Έχουμε την κυρία Μπουέρ από το Ίδρυμα Βεμός, ο κύριο ε, Στεφάν Φίρινγκ από την Αρμόδια Γενική τη Κομισιόν, ο κύριο. Ε, Φέργκισον από την ε, τη, τη διεύθυνση για τα φάρμακα και υπάρχει κάποιος άλλος υπάλληλος κομισιόν από την Γενική Διεύθυνση που αφορά την ε, έρευνα. Έχει το λόγο κυρία μου. Πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτούς που στις χώρε συμμετέχουν στις κλινικές δοκιμές. Αυτό γίνεται για νέα φάρμακα, οπότε και έχουμε και αυτές τις δοκιμές σε ανθρώπους. Ε, η έδρα του Ιδρυματός μας, του φορέα μας, είναι στις κάτω χώρες, Λατινική Αμερική, Αφρική, Ινδία, αναπτύσσουμε δραστηριότητα. Και οι εταίροι μας στις χώρες εκείνες είπαν ότι ανησυχούν για το στις αντιζόμενες χώρες ε, συνέχεια αυξάνονται αυτές οι κλινικές δοκιμές. Και συνήθως ε, γίνονται τέτοιες δοκιμές στην Ανατολική Ευρώπη, στην ε, Νότια Αμερική, Νότια, Νότια Αφρική, Νότια Αμερική και Ασία και δεν είμαι για αναπτυσσόμενες χώρες λέμε για κάποια φάρμακα που πηγαίνουν στη Δύση και όχι για κάποιες ασθένειε που υπάρχουν στην, σαν τις χώρες γιατί για τέτοιου φάρμακα δεν υπάρχουν επενδύσεις όπως για την ελληνοσία. εκτός Ένωση και είπα, να σας πω τι στοιχεία υπάρχουν από την Ευρωπαϊκό Χώρο των Φαρμάκων και στις χώρες που έχουμε κλινικές δοκιμές έχουμε κάποια φάρμακα τα οποία χρειάζονται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 20,3% το 2005 των ασθενών που συμμετείχαν σε τέτοιες δοκιμές για φάρμακα που θα πηγαίνουν στην Ευρώπη ήταν 20,3% εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα το 2008 ήδη μιλάμε για 33,9% περισσότερες χώρες που έγιναν αυτές οι δοχημές ήταν αναλυσόμενες χώρες ή αποδέκτες. το κέντρο έρευνας για την πολυεθνική συνεργασία λέει ότι έχουμε 18 έως 24.000 δοκιμές οι οποίες έγιναν σε κάποιες αναπτυσσόμενες φτωχές χώρες. Γιατί τώρα γίνονται όλο και περισσότερες δοκιμές σε αυτές τις χώρες. Πρώτα απ' όλα είναι πιο φθηνό να γίνουν εκεί αυτές οι δοκιμές. Επίσης λέει ότι θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει 200.000 δολάρια αν γίνει κανείς, κάνει κανείς σε τέτοιες χώρες τις ε, δοκιμές. Γιατί έχουμε κόστος 30.000 ανά, ανά άτομο, ανά δοκιμή, ενώ έχουμε 3.000. Ε, αν αντί για τις είπα γίνει αυτό σε αυτές τις χώρες. Επίση είναι και πιο εύκολα γενικότερα τα πράγματα, η διαδικασία, πιο εύκολα βρίσκει κανείς κόσμο, πρόθυμο να συμμετάσχει σε τέτοιες δοκιμές. Έχουμε και την εκθεσμένη μαγέση που έλεγε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε εάν κάνουμε πιο οικονομική διαδικασία πρόσληψη τατολογίας θα μπορούσαμε να, να, έχουμε τις οικονομίες 14 εκατομμύρια, γιατί στις, χώρες, στις ανεπτυγμένες χώρες μάλλον έχουμε ένα σωρό εγκρίσεις, επιτροπές, ιδιοντολογίες κλπ. να πρέπει να εξεταστεί δηλαδή επίσης το αν τα πειραματόζω έχουν εκτεθεί σε συναφή φάρμακα γιατί τότε τα αποτελέσματα θολώνουν. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτές τις αναδιωμένες αγορές και γι' αυτό και κατευθύνονται οι εταιρείε σε αυτές τις χώρες. Βεβαίω και έτσι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικά. Έχουμε στοιχεία που βοηθούν το ότι θεωρείται πολύ σημαντική ευκαιρία για την επιχειρηματική δραστηριότητα το να γίνονται αυτά τα, αυτές τις δοκιμές. Και στη Ρωσία το ίδιο. Ε, δύο δις, ένα δις είναι ο κύκλος εργασιών στην Ινδία και σύμφωνα με διάφορα ιδρύματα και εφημερίδες η Ινδική κυβέρνηση προσπαθεί να προσαρμόσει νομοθεσίες για λιγότερο αυστηρίο τόσο ώστε να γίνονται στη χώρα τους τέτοιες κλινικές δοκιμές. Επομένω, είναι επιχειρηματική ευκαιρία. Άμα θέλουν οι δύο επομένω οι ίδιοι να έρχονται οι δοκιμές χώρες. Γιατί εμείς να προβληματιζόμαστε. Προβληματιζόμαστε γιατί οι περισσότερες αντισόμενες χώρες δεν έχουν προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας, δεν έχουν ασφάλεια. Νοσοκομιακή περίθαλψη επομένως ε, πάνε στα πειράματα γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να έχουν θεραπεία και αγωγή φαρμακευτική. Δεν θεωρούμε πως λοιπόν, ότι έχουν επιλογή. Και εκτός αυτού τα μέτρα προστασίας των πειραματόζων δεν αποδίδουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Λειτουργούν καλά. Οι δε γιατροί που θα πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματα των ε, ασθενών είναι ίδιοι εμπλεγμένοι στην υπόθεση Μιλάμε για το ότι κάθε, ο καθένας που συμμετέχει ε, κοστίζει 13-15 χιλιάρικα, επομένως πώς, θα, πώς θα ενεργήσει ο γιατρός για να προστατεύσει τον ασθενή. στη Λατινική Αμερική καταγράφηκε ότι αυτοί που συμμετέσχουν είναι οι πιο αγράμματοι, φτωχοί και τελικά δεν καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που τους δίνονται. Ε, το βλέπουν σαν προϊστάμενό του τον ε, γιατρό. Για όμω λένε συμμετάσχουν, συμμετάσχουν, συμμετέχουν. Και έχουμε και θέσει επιτροπέ διοντολογία που υποτίθεται ότι είναι μέρος ενός μηχανισμού προστασίας και ούτε εκεί σε αυτές τις χώρες τα πράγματα δουλεύουν όπω θα έπρεπε. οι χωρέ αυτέ λένε οι μελέτες, δεν μπορούν να προστατεύσουν οι χώρε αυτέ οι σχετικέ επιτροπές τους. Ασθενείς που γίνονται πειραματόζωο. Ε. Υπάρχουν κάποιες ευθύνες γραμμές πάντως για την προστασία των όσων συμμετέχουν σαν πειραματόζωο. Έχουμε και μερικά κείμενα νομικά όπως η διακήρυξη του Ελσίνκη. Έχουμε κάποιες διακοινωτικές οδηγίες που παραπέμπουν εκεί το ειδικό δίκαιο για τέτοια πειράματα Όμως πολλές φορές παραβιάζονται οι διατάξεις αυτής της ε, διακήρυξης. Και έχουμε κάποιες δοκιμές για φάρμακα που θα πήγαιναν μετά στην Ευρώπη, αλλά δοκιμάστηκαν στην Ινδία. Ήταν κάποιο φάρμακο που αφορούσε κάποιους ε, καρκινοπαθείς με ε, καρκίνο στο στήθος και τελικά ήταν τόσο, τόσο ακριβό αυτό το φάρμακο που δεν μπορούσαν να το αγοράσουν οι καρκινοπαθείς. Ε, δεν πρέπει να καταβάλουν περίπου 1000 ευρώ το μήνα. Ε, οι δηλαδή, επόμενε αυτοί κάνουν τις δοκιμές, είναι πειραματόζω και δεν έχουν το και τα λεφτά μετά να αγοράσουν το φάρμακο. Επίσης, ε, άλλο παράδειγμα, ε, έχουμε ένα φάρμακο κεφαλική διαταραχή, διανοητική διαταραχή. Ε, κάποιοι από αυτούς που συμμετέσχουν ήταν ασθενείς, είχαν πρόβλημα, τους δώσανε από το φάρμακο και είπε μετά η εταιρεία ότι οι επιτροπές διοντολογίας δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους τέτοιου είδου πειράματα με αυτή τη μέθοδο. Βλέπω ότι έχω δύο λεπτά μόνο και πρέπει να βιαστώ. Αλλά βλέπετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συχνά απευθύνει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει γίνει μία συνάντηση εμπειρογνωμόνων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και την φαρμακοβιομηχανία και η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει ε, το θέμα. Η σχετική μελέτη ε, δημοσιεύθηκε πέρυσι, διατυπώνει ορισμένες συστάσεις είτε για το ρυθμιστικό πλαίσιο είτε ε, για νέες μεθόδους και θεωρούμε ότι όσον αφορά την ισχύουσα νομοθεσία έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο κάθε ευκαιρία να προστατεύσουμε τις, τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις δοκιμές αυτές της υποανάπτυξη χώρες διότι για να μπορέσει να υπάρξει μία άδεια εμπορίας για κάποιο φάρμακο πρέπει να υπάρχει σεβασμός της διακήρυξης του Ελσίνκη και των κατευθυντηρίων ε, γραμμών ε, και εάν ε, αυτά δεν έχουν εφαρμοστεί δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα. Υπάρχει το Ευρω... ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων που εξετάζει το θέμα αυτό αλλά εμείς θεωρούμε ότι όσον αφορά την αγωγή μετά από την, τις δοκιμές και με τα εικονικά φάρμακα δεν έχει προχωρήσει κανείς τόσο αποτελεσματικά και ε, θεωρούμε σαν καταναλωτές των φαρμάκων που δοκιμάζονται στις υποανάπτυξη χώρες ότι θα έπρεπε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας προς τα άτομα αυτά που χρησιμοποιούνται σαν πειραματόζωμα. Ε, ε, τόσο Ευχαριστώ. Ξέρετε όμως ότι το πρόβλημα του χρόνου υπάρχει πάντοτε σε εμά, Ο κύριος Στέφαν Φιούρινγκ έχει τώρα το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Στέφαν Φούρινγκ. Ε, εργάζομαι στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών και ε, παρακολουθώ το φάκελο αυτό. Καταρχήν σας ευχαριστούμε που ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό και μας απασχολεί πάρα πολύ και το έχουμε περιλάβει και σε μία ε, ανοιχτή διαβούλευση για μία μία αξιολόγηση επιπτώσεων σχετικά με τις ε, ε, κλινικές δοκιμές. Υπάρχει βέβαια η έκθεση αυτή την οποία έχετε καταρτήσει και την οποία επίσης ε, έχουμε επεξεργαστεί και έχω να πω τέσσερα πράγματα στο σημείο αυτό. Καταρχήν ε, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι λανθασμένο να πει κανείς ότι οι κλινικές μελέτες εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη δοκιμάζονται μαζικά στις υποανάπτυξη χώρες. Δεν συμφωνούμε με τους αριθμούς οι οποίοι ανεφέρθησαν διότι οι αριθμοί που έχουμε εμείς μας δείχνουν μια διαφορετική εικόνα όσον αφορά τις κλινικές μελέτες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων από το 2005 έως το 2008 10% ήταν από την Ασία και 10% από την Νότιο Αμερική αλλά σχεδόν κανένα, καμία δοκιμή δεν έγινε στην Αφρική. Επίσης δεν είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που ελέγχει lengthy the majority of uh, clinical uh, trials uh, συμβαίνει στις υποανάπτυξη χώρα, δηλαδή η πλειοψηφία ε, και ότι υπάρχουν πλέον των 20.000 κλινικών δοκιμών που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αφρική γιατί ε, στην Ευρώπη έχουμε τυσίως περίπου 5.500 κλινικές δοκιμές το χρόνο δηλαδή δεν υπάρχει καμία μετακίνηση της της από την Ευρώπη προς τις υποανάπτυξη χώρες. Όσον αφορά την έκθεση, οι κλινικές μελέτες προς τις τρίτες χώρες είναι μία πρόκληση αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι εκ προημίου η ποιότητα των κλινικών αυτών δοκιμών είναι χειρότερη και ότι υπάρχει κλινικό dumping από την άποψή μας ε, αυτό δεν συμβαίνει γενικά. Θα πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε τα υπάρχοντα στοιχεία και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις ε, ε, τις επενδύσεις. Επίσης πρέπει να παρακολουθεί κανείς το θέμα διότι βεβαίως οι κλινικές δοκιμές είναι όλο και πιο γενικευμένες λαμβάνουν χώρα και σε τρίτες χώρες, σε πιο φτωχές τρίτες χώρες για πολλούς και διάφορους λόγους όχι πάντοτε αναγκαστικά γιατί είναι πιο φτηνά ή πιο γρήγορα αλλά για ρυθμιστικούς λόγους διότι ορισμένες τρίτες χώρες απαιτούν να έχει γίνει μία δοκιμή στο κράτος τους για να εγκρίνουν ένα φάρμακο. Οπότε πρέπει και το στοιχείο αυτό να ληφθεί υπόψη. Και τέλος, το τελευταίο στοιχείο, όπως ελέγχθη, συμφωνούμε ότι πρέπει να υπαγρυπνούμε στο θέμα αυτό. Βεβαίως προσκρούομαι ε, στα θεσμικά μας όρια. Υπάρχει και ένα θέμα της δικαιοδοσίας και το καλύτερο στοιχείο που έχουμε είναι η άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάκου στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να υπάρχουν κλινικές μελέτες είτε σε εθνικό επίπεδο είτε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Όταν λοιπόν ε, φτάνουμε σε αυτό το σημείο της ε, ε, διασύνδεσης δικαιοδοσίας μπορούμε να κάνουμε ελέγχους και να προσφύγουμε σε επί, σε ελέγχους και η Επιτροπή έχει αναλάβει σε αυτό το θέμα πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σουάινι της Γενικής Διεύθυνσης Φαρμάκων για πέντε λεπτά. Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Σουίνι Είμαι υπεύθυνο της συμμορφώσεω και των ε, ε, επιθεωρήσεων ε, στο γενικό, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Το θέμα αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ. Παρακολουθούμε την πρόοδο και τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία χρόνια έχουμε συνήθως, έχουμε επίσης εξετάσει τις μελέτες οι οποίες λαμβάνουν κάνουν χώρα στη Βόρειο Αμερική και στην Ευρώπη και έχουμε καταρτήσει μία έκθεση για την περίπτωση, ε, περίοδο 2005-2008 θα προσθέσουμε ως ονούπο τα στοιχεία για το 2009. Κατόπιν λοιπόν του εγγράφου το οποίο είχαμε δημοσιεύσει το 2008 έχουμε καταρτήσει μία ομάδα εργασίες που αποτελούνται από εκπροσώπους της ομάδος παιδιατρικής, της ομάδος ε, φαρμάκων για ανθρώπους ε, και άλλων και ετοιμάζουμε ένα ε, έγγραφο προς ε, εξέταση για να εντοπίσουμε ε, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουμε να ε, κάνουμε μελέτες στις διάφορες χώρες και να μπορέσουμε να περιλάβουμε τις κλινικές μελέτες και μελέτες με φάρμακα και εικονικά φάρμακα συγκρίσεις και τα λοιπά και επίσης να μπορέσουμε να δώσουμε καθοδήγηση και συμβουλές. Αυτά τα δύο βήματα θα εξασφαλίσουν ότι θα προεξοφλήσουμε ότι οι κλινικές μελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την εφαρμογή του φαρμάκου. Θέλουμε λοιπόν να έχουν γίνει αυτές οι κλινικές μελέτες και αυτό το οποίο να βάλουμε υπόψη μας όταν εξετάζουμε την κατάσταση της αγοράς και τα ηθικά πρότυπα είναι να εξετάσουμε το θέμα των επιθεωρήσεων και, ε, των, ε, και το αξιολογήσεως, της διαφάνειας για να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζονται οι ηθικές προδιαγραφές και τέλος προσπαθούμε να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία διότι όπως ελέγχθη εν τρίτον των μελετών γίνονται στην Ευρώπη, εν τρίτον στην Βόρειο Αμερική και εν τρίτον στον υπόλοιπο κόσμο αλλά στις στατηγικές μας μόνο οι ουσιαστικές μελέτες 33.000 λαμβάνονται υπόψη οπότε δεν παρακολουθούμε τα πάντα. Αυτό που είναι βασικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό στις χώρες ε, το οποίο να είναι ισχυρό και να στηρίζεται ε, ε, τα σωστά μέτρα κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ηθική, ηθικά ορθή διεξαγωγή των μελετών αυτών και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε επιθεωρητές αλλά και πρόπερση και όχι μόνο από την Ευρώπη και τα νέα κράτη-μέλη αλλά από την Ινδία, από την Ασία, από την Αφρική, από την Νότιο Αφρική και αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί με τους εταίρους μας και από την Βόρειο Αμερική για να εξασφαλίσουμε ότι οι σωστές μελέτες γίνονται όπου και όπως πρέπει. Το Σεπτέμβριο εφέτος μετά από την δημοσίευση του εγγράφου που προανέφερα θα υπάρξει μία ενημέρωση του εγγράφου το δεύτερο εξάμεινο. Ευχαριστώ και τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Ρωμάρης της Γενικής Διευθύνσεως Μελετών. Οι περισσότερες μελέτες γίνονται στις ανάπτυξη χώρες και εκεί χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατόπιν ε, πρωτοβουλίας κοινή από το Συμβούλιο και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να, ε, να υπάρξουν κλινικές μελέτες για μικροβιοκτώνα, ε, εμβόλια και άλλα φάρμακα και στην Αφρική. Ακολουθούμε όμως τα ε, ήδη υψηλά πρότυπα ηθικής τα οποία ισχύουν και στην Ευρώπη και παρακολουθούμε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούμε. Άλλωστε για να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδοτούμε και έρευνες για τα ηθικές προδιαγραφές και εξετάζουμε τις ε, εθνικές και διεθνείς πτυχές για να ξέρουμε ότι εφαρμόζονται και ε, χρηματοδοτούμε και ένα ε, φόρουμ εμβολίων στην Αφρική συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και χρηματοδοτούμε δράσεις στην Αφρική μέσω διαφόρων οδών οργανώνουμε και σειρές μαθημάτων και εργαστήρια. Στα 7 χρόνια που υπάρχει ο οργανισμός μας έχει χρηματοδοτήσει μία σειρά προγραμμάτων για ένα ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2010 ε, υποβάλαμε νέες προτάσεις για 75 εκατομμύρια ευρώ για να δημιουργήσουμε τέτοια συμβούλια στην ε, υποσαχάριο Αφρική. Πρέπει να πούμε ότι όλα τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε στην Αφρική ε, έχουν την ίδια μορφή με τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούμε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 ή έχουμε πρόβλημα ή πολύ υπερβάλλουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί ή μήπως υπερβάλλουμε για κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μικρό πρόβλημα. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο πρώτος ομιλητής, η πρώτη ομιλήτρια μάτων, ουσιαστικά θέλει να μας πει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες κάνουν τεστ σε ανεψόμενες χώρες και ιδιαίτερα στην Ινδία σε φάρμακα που δεν θα κάνουν τεστ στην Ευρώπη εκτός αν ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Η πρώτη ομιλήτρια μας λέει ότι οι ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες κάνουν τεστ για φάρμακα σε άτομα σε ανεψόμενες χώρες και στην Ενβία που δεν θα, για τα οποία δεν θα κάνουν κλινικό έλεγχο σε Ευρωπαίους επειδή το φάρμακο αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτό μας είπατε. Το κόστος είναι μηχανισμός αγοράς. Δεν θα μιλήσουμε για την αγορά. Αν όμως ο ισχυρισμό σας είναι ότι ορισμένα φάρμακα που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνα αν γίνει τεστ γίνεται τεστ στις αναπτυσσόμενες χώρες διότι η ζωή ενό προσώπου στην αναπτυσσόμενη χώρα δεν είναι τόσο σημαντική όσο η ζωή ενό Ευρωπαίου. Τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχουν αποδείξει ότι οι φάρμακοβιομηχανίε κάνουν τεστ κλινικέ δοκιμέ, τεστ πειραματικά φάρμακα σε ένα άτομα των αναπτυσσόμενων χωρών που δεν θα τους περνούσε καν από το μυαλό να δοκιμάσουν να κάνουν τέτοιο τεστ σε Ευρωπαίους. Χρειάζομαι απάντηση σε αυτό. Δεύτερον, αν είναι θέμα εποπτείας, εμείς έχουμε αρκετούς πόρους ώστε να μπορούμε να υποπτεύουμε τα τεστ που γίνονται στις αναπτυσσόμενες χώρες από ευρωπαϊκές εταιρείε. Τρίτη ερώτηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, η κυβέρνηση εννοώ, τι κάνουν για τις Αμερικάνικες εταιρείε όταν κάνουν ας πούμε τεστ στη Λατινική Αμερική. Συνεργαζόμαστε με αυτούς, έχουμε υιοθετήσει τις μεθόδους τους, άριστες μεθόδους κλπ. Έχουμε διαφορετικό σύνολο προδιαγραφών για μας. Η κυρία Σαργεντίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις προς την Κομισιόν. Ακούγοντας τη συζήτηση και επειδή ο κύριος Ντέβα έθεσε ένα πολύ ηθικό ερώτημα. Το ερώτημα αυτοί που κάνουν τα τεστ για μας στις αναπτυσσόμενες χώρες μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακα αυτά αν χρειαστεί ή όχι. Γιατί μιλάμε για ακριβά φάρμακα και αφού γίνει ο έλεγχος μετά τα άτομα δεν έχουν χρήματα για να συνεχίσουν τη θεραπεία Συχνά η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι όχι. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν τώρα να μας πει στο μέλλον μπορεί να μας διασφαλίσει ότι ο οργανισμός φαρμάκο θα ελέγχει πριν κυκλοφορήσει ένα φάρμακο στην Ευρώπη για τη δήλωση του Ελσίνκη, αν τηρήθηκε η δήλωση του Ελσίνκη, Άλλη ερώτηση. Η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να αλλάξει τους κανόνες για, για τα τεστ πλασίμπο σε τρίτες χώρες. Στην Ευρώπη μια σοβαρή ασθένεια δεν μπορούμε να πούμε αυτό ε, είναι ένα φάρμακο για το οποίο έγινε τεστ, το άλλο είναι πλασίμπο. Σε χώρες όπως η Ινδία αυτό συμβαίνει όμως. Δηλαδή οι φαρμακοβιομηχανίες πάνε εκεί γιατί αυτού του είδους τα τεστ δεν τους επιτρέπονται να τα κάνουν στην Ευρώπη, από ό,τι ξέρω. Αυτά τα φάρμακα δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά αν έχουν περάσει τέτοιου είδους τεστ, αν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Έρευνα λοιπόν για τον έλεγχο των πλασίμπο, των εικονικών φαρμάκων. Μετά, αν επιτρεπεί να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο στην Ευρώπη έχοντας υποστεί τεστ σε τρίτη χώρα. Να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε οι χώρες στις τρίτη χώρες και αυτοί να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο αυτό. Διότι αυτό το ηθικό ερώτημα αφορά και την τιμή και το ποια ζωή αξίζει περισσότερο εδώ στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες. Αυτό ισχύει όταν μιλάμε για τον κλινικό έλεγχο των φαρμάκων. Γκέρενς. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Αν ε, έχουμε κατάχρηση του συστήματος, το ερώτημα είναι ποιο νομικό καθεστώς ισχύει. Το ευρωπαϊκό των κρατών μελών αν ισχύει αυστηρά Ακόμα και αν οι κλινικές ε, δοκιμές γίνονται σε τρίτες χώρες, αν διαπιστωθεί μια κατάχρηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ερώτημα είναι ισχύει η δική μας νομοθεσία. Αν ναι, αυτό θα ήταν αποτρεπτικό σε σχέση με τις ενδεχόμενες καταχρήσεις, κατάχρηση μάλλον του συστήματος. Δεύτερον, δεν μπορούμε να απομονώσουμε τις κλινικές δοκιμές από την πρόσβαση στα φάρμακα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και συμφωνώ με αυτό που είπε η κυρία Σαρζεντίνη. Λέμε, ένα τρίτο των κλινικών δοκιμών γίνεται στην Ευρώπη, το υπόλοιπο γίνεται στη Βόρεια Αμερική, υποθέτω το υπόλοιπο τρίτο γίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο καταμερισμός των φαρμάκων όμως στον κόσμο δεν ανταποκρίνει σε αυτού του είδους την διαίρεση. Άρα μπορεί να μην έχουμε ενδεχομένω ατομικά ηθικό πρόβλημα όσον αφορά την εφαρμογή των κλινικών ελέγχων. Έχουμε ηθικό πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Έπειτα αυτό συνδέεται με την έρευνα για τα φάρμακα. Θα ήθελα να ακούσουμε δύο λόγια για τα δημόσια κονδύλια που πάνε στην έρευνα για τις τροπικές ασθένειες και ασθένειες που δεν είναι πάρα πολύ γνωστές που όμως είναι χαρακτηριστικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι για τις χώρες του Βορρά. Χρειαζόμαστε απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα προκειμένου να πούμε αν η πολιτική μας μπορεί να χαρακτηριστεί ηθική σε θέμα στην, όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Σας θυμίζω ότι η ασύμετρη θεραπεία στο θέμα αυτό οδήγησε την Ινδονησία να αρνηθεί να δώσει στελέχη για επεξεργασία εμβολίων, στελέχη ιού ενώ, προκειμένου να γίνουν εμβόλια κατά των ασθενειών αυτών. Μπορεί κατά περίπτωση να μην υπάρξουν ηθικά, να μην υπάρχουν ηθικά προβλήματα, υπάρχει όμως ένα ουσιώδες ηθικό πρόβλημα που αφορά το σύνολο και αφορά ουσιαστικά το θέμα πρόσβασης στα φάρμακα για τα 4 πέμπτου του πληθυσμού της γης. Η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Μια ερώτησή μου προς τον κύριο Μπέρμπουρ, δεν ξέρω πώς προφέρει το όνομα. Αναφερθήκατε στη δήλωση του Ελσίνκη σε σχέση με τον έλεγχο και είπατε ότι υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα στην εφαρμογή γιατί δεν εφαρμόζεται η διακήρυξη του Ελσίνκη και ποιος είναι ο ρόλος σας. Ο κύριος Σαλόμ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας είναι ένα από τα πρωτεύοντα δικαιώματα του ανθρώπου και της αναγνώρισης της ισότητας των ανθρώπων. Ακούσαμε νούμερα και ποσοστά και αναλύσεις διαφορετικές ανάλογα με το αν μιλούσε εμπειρογνώμονες ή εκπρόσωπος κομισιών. Υπήρξε όμως ένα κοινό σημείο κατά τη γνώμη μου παραδοχή ότι η Ένωση έχει νομοθεσία και μηχανισμούς επαρκής για να ρυθμίζει αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό. Και ρωτώ την Κομισιόν. Συμφωνεί ή όχι με αυτό που είπε η εκπρόσωπος του Ιδρύματος για το ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν τηρείται επαρκώς ή αυστηρά. Και αν η Κομισιόν δεν έχει σήμερα χρόνο να δώσει μια εκτενή απάντηση στο ερώτημα, τουλάχιστον ας στείλει στην Επιτροπή μας μια έκθεση για το βαθμό εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πρόεδρος. Το λόγο στην κυρία Ντενμπουέρ του Ιδρύματος Βέμος για να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν και επίσης σας έκοψα κάπως απότομα πριν θα σας δώσω λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι θα δώσω στους τρεις εκπροσώπους της Κομισιόν. Ευχαριστώ για τη γενοδορία σας κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, γι' αυτό που είπε ο κύριος Φύρινγκ της Κομισιόν. Εγώ δεν είπα ότι τα περισσότερα τεστ γίνονται εκτός της Ένωσης και των Πολιτειών. Είπα ότι οι περισσότεροι ασθενείς που παίρνουν μέρος στα τεστ αυτά εκτός της Ένωσης και των Πολιτειών είναι από αναπτυσσόμενες χώρες. Από το 1 τρίτο που γίνεται εκτός Ευρώπης και Αμερικής είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και οι περισσότερες χώρες είναι στον κατάλογο των δικαιούχων του ODA. Αυτό εννοούσα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε ευθύ εξ αρχής. Δεύτερο, εσείς επίσης αναφερθήκατε στο ότι οι κλινικές δοκιμές γίνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν σημαίνει ότι είναι ίσονος σημασίας και ποιότητας. Ωστόσο, η έρευνα μας δείχνει ότι η ποιότητα των μηχανισμών ελέγχου στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως είπα, επιτροπές ηθικής κλπ, δεν είναι επαρκής. Αναφέρθηκα σε μια επισκόπηση για το λατινικό δίκτυο ηθικής. Πολλές από τις επιτροπές ηθικής δεν έχουν προσωπικό αρκετό, δεν έχουν καλή εκπαίδευση. Υπάρχει ένα διορθωτικό πρόβλημα. Χαίρομαι για το ότι ο κύριος Σουίνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου αναφέρθηκε στο ότι η Ένωση παίρνει πρωτοβουλίες για να ενισχυθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό είναι σημαντικό βήμα και είναι ουσιαστικά τελικά θα είναι η λύση για τα ηθικά τεστ. Έχουμε περισσότερους ελέγχους, αλλά όπως ο κύριος Φίνη, δεν είναι αυτή η λύση γιατί γίνονται πάρα πολλέ κλινικές δοκιμές και είναι αδύνατο να τις καλύψουμε όλους, όλες τα τεστ αυτά με ελέγχους. Και έρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Μπέρμαν. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε συνέντευξη με οι διάφορους φορείς φαρμάκων στην Ένωση και τους ρωτούσαμε ελέγχεται αν ένα φάρμακο ελέγχθηκε με βάση αρχές της διακήρυξης του Ελσίνκη και οι περισσότεροι απάντησαν όχι. Μερικοί είπαν ότι αυτό δεν είναι ακόμα στο σύστημά μας. Ε, κοιτάμε την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, αλλά όχι το ηθικό σκέλος, ελάχιστα. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να γίνονται ηθικοί έλεγχοι όσο πιο σύντομα γίνεται στη φάση των κλινικών δοκιμών. Και όχι μόνο όταν το φάρμακο μπαίνει στην αγορά. Θα ήταν βελτίωση αν γινόταν τέτοιου είδους έλεγχη. Ως τα φάρμακα αν συμμορφώνονται δηλαδή με τη διακήρυξη του Ελσίνκη. Σοβαρά. Πριν τους δοθεί η έγκριση να μπουν στο κύκλωμα της αγοράς. Στην ερωτήσει του κυρίου Ντέβα δεν κοιτάμε μόνο τις ευρωπαϊκές εταιρείες, κοιτάμε πολυεθνικές επιχειρήσεις που κάνουν κλινικές δοκιμές σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έδωσα ένα παράδειγμα της Άστρα η οποία παραδέχτηκε ότι έκανε έναν έλεγχο πλασίμπο εικονικών φαρμάκων στην Ινδία, γιατί υπάρχει μια... Η, η, Επιτροπή Ηθικής στην Ευρώπη αυτό δεν θα το επέτρεπε ποτέ. Ελπίζω να απάντησα. Ντέβα. Όχι, όχι. Μια δοκιμή. Αφ, αφήστε καλύτερα την κυρία Μπόρ να τελειώσει και μετά. Η κυρία Μπόρ συνεχίζει. Το κατά πόσο είναι διακήρυξη του Ελσίνκη γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά. Αυτό οφείλει στο ότι δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Θεωρούμε ότι θα ήταν πολύ σημαντικό βήμα όπως το ζήτησαν ε, οι ευρωβουλευτές που μίλησαν να γίνει αυτό παραδείγματο χάρη η τιμή των φαρμάκων να είναι χαμηλότερη για χώρες που παίρνουν μέρος στα τεστ. Αν μπορούσε να γίνει έλεγχος πριν δοθεί έγκριση εμπορίας του φαρμάκου. Νομίζω ότι απάντησε στις περισσότερες ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. λίγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Στεφάν Φέρινγκ και στους άλλους δύο εκπροσώπους της Κομισιόν αν θέλετε για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι ερωτούντες όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και αν επαρκεί. Είναι σαφές αυτή τη στιγμή κάθε μελέτη η οποία κατατίθεται στην Ευρώπη σε σχέση με την ε, άδεια κυκλοφορίας ενός φαρμάτου πρέπει να συνάδει με τις αρχές της κλινικής πρακτικής και ε, σε αυτό βασιζόμαστε και στις διεθνείς συμφωνίες. Πιο ουσιαστικό είναι το θέμα της ουσιαστικής εφαρμογής της ε, αφηρημένης νομοθεσίας και είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ. Όσον αφορά ε, την, το, την επαλήθευση των κατατεθειμένων στοιχείων σε σχέση με την ε, συμμόρφωση προς τις ηθικές αρχές είναι κάτι ε, το οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ρυθμιστικά μέτρα τα οποία τώρα μελετούμε. Καταρχήν είναι η διαφάνεια. Όσο πιο διάφανη είναι η κλινική μελέτη ε, την τρίτη χώρα τόσο πιο έγκαιρα μπορούμε να προβούμε σε κλινικές επαληθεύσεις και πιέζουμε τους επιθεωρητές να ε, εξασφαλίσουν ότι οι μέθοδοι που εφαρμόζουν συνάδουν με τις ε, εθνικές ηθικές μεθόδους. Και ένα τελευταίο θέμα σχετικά με τις ε, επιθεωρήσεις δεν είναι δυνατόν ε, για όλα τα ε, νοσοκομεία και για όλα τα Ινστιτούτα να προβαίνουμε σε ελέγχους γιατί υπάρχουν εκατοντάδες ε, χιλιάδες ενδεχομένως ιδρυμάτων για μία κλινική μελέτη και γι' αυτό πρέπει να αναπτύξουμε το δυναμικό και χαιρόμαστε ότι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι ερευνητικές αρχές και ε, ο σχετικός οργανισμός. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ και πάλι που μας δώσατε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Thank you. Um, just to pick on Ευχαριστώ. Θέλω να αναφερθώ ε, και να σχολιάσω ένα-δύο θέματα συνεργαζόμαστε με την FDN στις Ηνωμένε Πολιτείε και με άλλους οργανισμούς οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στην ε, ε, ομάδα εργασίας ε, επιθεωρητών πράγμα το οποίο θα γίνει και στην ομάδα Αφρικής ε, και Ασίας και σε αυτό το θέμα όπως και σε άλλα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι ευθύνες κατανέμονται σωστά και ότι δεν παρακολουθούμε μόνο ένα χώρο αλλά όλους τους χώρους για να υπάρχει σωστή ε, επιτήρηση όλων των δοκιμών και αυτό σε, σχέση, ε, σε, συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης με την ε, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και όποιου συνεργάζεται με αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά τις, το σχεδιασμό των μελετών, τον οποίο έχουμε παρακολουθήσει ε, και θα συνεχίσουμε να ε, παρακολουθούμε. Ε, θα προσκαλέσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους από όλες τις χώρες να επανέλθουν στο θέμα αυτό. Επίσης, όπως ανεφέρθη προηγουμένως, μέχρι μέσω του άρθρου 58 προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τις ε, ε, ε, άδειες κυκλοφορίες και για άλλα φάρμακα όπως είναι η ελονοσία, η φυματίωση δηλαδή θέματα τα οποία θίγει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πιστεύουμε ότι η διακήρυξη του Ελσίνκη και σχετικά με τις κλινικές μελέτες συμπληρώνεται ε, διότι ε, αναφέρεται στις πιο πρακτικές πτυχές των κλινικών μελετών. Είναι δύο θέματα τα οποία πρέπει να συνδυάσουμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις μεθόδους μας, να βελτιώσουμε την επιμόρφωση που προσφέρουμε για την εφαρμογή των δοκιμών. Ευχαριστώ κυρία ε, Πρόεδρε. Ε, θέλω να επανέλθω στο θέμα των τροπικών ασθενειών διότι ε, υπάρχει μία, ένα πρόγραμμα για τις τροπικές ασθένειες. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζουμε ένα δεύτερο τέτοιο πρόγραμμα. Ελπίζουμε από το 2010 να δημιουργηθεί μη ένα τρίτο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να έχουμε μία πιο βελτιωμένη εφαρμογή μετά το 2010. Δεν μου απάντησε κανείς από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους ελέγχους οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί σε πιο ποσοστό των ε, ε, δοκιμών. Όσον αφορά τις δοκιμές σε σχέση με το με το θέμα αυτό έχουν σχέση με την επιτήρηση της GCP διότι όπως ξέρετε ένα πολύ μικρό ποσοστό μόνο από τις δοκιμές μπορεί να επιθεωρηθεί και πρόκειται για μία δειγματοληψία για να δούμε και τα συστήματα και της χώρας και τις επιχειρήσεις για να δούμε αν γίνονται σωστά οι δοκιμές. Το 2009 έγιναν 58 τέτοιες μελέτες και ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί βαθμιαία και πάνω από τις μισές ε, δοκιμές γίνονται σε τρίτες χώρες. Προσπαθούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε όταν κάνουμε τις επιθεωρήσεις ότι θα αυξήσουμε ε, το ποσοστό των χωρών στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική όπου προβαίνουμε σε ελέγχους των δοκιμών. Ε, έχουμε μία πρώτη έκθεση ε, το 2005 έως 2008 και ε, θα δημοσιεύσουμε ως ο Νούπο την αναθεωρημένη προέκταση στο 2009. Ε, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δύο ευρωβουλευτές ακόμη δεν έχουν λάβει απάντηση και θέλουν μια ερώτηση ε, διευκαινιστική να κάνουν. Η κυρία Σαργεντίνη και μετά ο κύριος Ντέβα. Ε, ευχαριστώ. Δεν πρόκειται για διευκρινιστική ερώτηση. Θα ξανακάνω την ίδια ερώτηση για να μου δώσουν μία απάντηση. Γιατί βλέπω ότι ξεδιαλέγουν τις ερωτήσεις και απαντούν κατά βούληση. Ε, ρωτάω λοιπόν και πάλι. Επιτροπή, είναι δυνατόν στο μέλλον να ελέγχουμε όντως εάν η διακήρυξη ε, του Ελσίνκη έχει εφαρμοστεί προτού δώσουμε πρόσβαση στα φάρμακα και οι μελέτες που γίνονται στις ε, τρίτες χώρες να μην γίνονται με την ε, μέθοδο των εικονικών φαρμάκων που δεν είναι δεκτή στην Ευρώπη ε, να έχουμε πρόσβαση στα φάρμακα και να ε, εξασφαλίσουμε ότι τρίτες χώρες που χρησιμοποιούνται ε, σαν χώρος για τις δοκιμές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που δοκιμάστηκαν στην επικράτειά τους. Θέλω να επανέλθω στο ίμιση της ερωτήσεως το οποίο είχα κάνει πριν. Ε, ξέρω τι κάνουμε για τα εικονικά φάρμακα, αλλά αυτό που ήθελα να διευκρινίσω είναι, είναι προφανές ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, μελετούν φάρμακα στις αναρτησόμενες χώρες τα οποία δεν θα χρησιμοποιούσαν για δοκιμές σε Ευρωπαίους ασθενείς. Ο κύριος Γκιόρενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξέρω εάν οι παρεκτροπές παραδείγματος χάρη μιας γαλλικής εταιρείας στις ε, κλινικές δοκιμές σε μια υποανάπτυξη χώρα θα τιμωρηθούν σύμφωνα με την γαλλική νομοθεσία ή με την νομοθεσία του υποανάπτυξη κράτους. Και ε, τέλος ο κύριος Μπέρμε. Όχι, τέλειωσε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επρόκειτο για ερωτήσεις προς την Επιτροπή αντιλαμβάνομαι ότι δεν ικανοποιήθηκαν οι ε, βουλευτές ε, ότι ε, υπάρχουν σωστές μελέτες προτού δοθεί η έγκριση κυκλοφορίας στην αγορά του φαρμάκου και θα ήθελα η Επιτροπή να μας απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, ήδη τώρα κάθε μελέτη η οποία υποβάλλεται ελέγχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ε, την, ε, ε, τα συμπεφωνημένα. Επίσης, εάν μία μελέτη δεν συμμορφώνεται ως προς τις ηθικές επιταγές, θα πρέπει να απορριφθεί η, η έγκριση και να μην της δοθεί η δυνατότητα, δεν να μην δοθεί δυνατότητα να ε, ισχύσει αυτό το φάρμακο. Επίσης όσον αφορά το follow-up treatment, η παρακολούθηση, η, ε, η αγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τοποθετούν ε, βέβαια πολλά προβλήματα, προκύπτουν πολλά προβλήματα, και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί ε, την ε, ομάδα η οποία το επεξεργάζεται και θα υπάρξει ε, μία απάντηση μέχρι το Σεπτέμβριο εφέτος. Επίσης, αν ένα φάρμακο δοκιμαστεί κλινικός από μια γαλλική εταιρεία σε μια, μια τρίτη χώρα και παραβιάσει την νομοθεσία του τρίτου κράτους θα διωχτεί σύμφωνα με την νομοθεσία του τρίτου κράτους και όχι της Γαλλίας αλλά εάν δοθούν αυτά τα στοιχεία από την εταιρεία για την αδειοδότηση του φαρμάκου θα πρέπει να συμμορφώνεται και με την εθνική νομοθεσία διότι διαφορετικά θα μπορέσει κανείς να απορρίψει τα στοιχεία αυτά. Λοιπόν, ας μείνει εδώ η συζήτηση και θα έλεγα η Επιτροπή Ανάπτυξης να συνεχίσει να παρακολουθεί ε, εκ του ε, το πόσο προχωράει το θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα Προχωράμε ε, στο σημείο 10 γιατί είμαστε λιγάκι άτακτοι λόγω της ε, αλλαγής που κάναμε στο πρόγραμμα. Μιλάμε για την επίτευξη πρόοδου όσον αφορά την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ενδιάμεση αναθεώρηση για την προετοιμασία της συνεδρίας υψηλού επίπεδου το Σεπτέμβριο 2010, όπου η συνεδρία θα γίνει στη Νέα Υόρκη για να αξιολογήσει τι τα πρόοδους που επετεύχθησαν, λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε μόνο πέντε χρόνια πριν από την καταληκτική ημερομηνία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μία κοινή ευρωπαϊκή θέση εν ώψη αυτής της συνεδριάσεως. Θα πρέπει μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε καταλήξει σε αυτή την κοινή ε, φιλόδοξη θέση και ο κύριος Κάσμαν προετοιμάζει ε, μία, ε, ένα ψήφισμα. Σας έχει ήδη διανύμει ένα έγγραφο εργασίας και έχουμε σήμερα καλέσει τρεις εμπειρογνώμονες, την κυρία Φρονσουάζ Μωρό, ε, διευθύντρια του τμήματος στην Επιτροπή που ευθύνεται για την κατάρτιση της προτάσεως σχετικά με τους στόχους της χιλιατηρίδας που θα υπάρξει στο έγγραφο της Ανοίξεως και ε, ένα και δύο ακόμη ε, εμπειρογνώμονες ένα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και ένα από την υπεύθυνη διεύθυνση. Καταρχήν έχει το λόγο ο κύριος Σκάσουμεν για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ βασικό να κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατό να εξασφαλίσουμε ότι το ψήφισμα αυτό θα είναι έτοιμο για την Ολομέλεια του Ιουνίου για να μπορέσει να επηρεάσει την κατάσταση. Καθότι μιλάμε τόσο πολύ για τη φτώχεια και τα προβλήματα του κόσμου και νομίζω ότι όσο περισσότερο συζητάμε τόσο λιγότερο πλησιάζουμε μία λύση για να υπάρξει δράση. Και το λέω αυτό διότι ε, είναι καλό να μπορεί κανείς να αναλάβει αυτή την ενέργεια εν ονόματι ε, του Κοινοβουλίου και ε, θα ήθελα ήθελα να μιλώ εγώ λιγότερα, να με ακούν περισσότερο για να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα επιτύχει πραγματική πρόοδο. Είχαμε μεγάλες προσδοκίες από την Κοπεχάγη και αποτύχαμε. Η αποτυχία αποτύχαμε, η αποτυχία όμως τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο δεν είναι ανεκτή κάναμε μία μία υπόσχεση ε, εις ε, τους φτωχούς ότι πράγματα τα οποία θεωρούμε ως ε, προεξοφλημένα όπως πρόσβαση στην υγεία, πρόσβαση σε καλή διατροφή, στο νερό και σε εκπαίδευση θα υπάρξει και για αυτούς. Κάναμε ε, λοιπόν ε, ε, υποσχέσεις τις οποίες πρέπει τώρα να σεβαστούμε και να προχωρήσουμε. Δεν θα πω λοιπόν τίποτα παραπάνω, θα ακούσω τους εμπειρογνώμονες, διάβασα το έγγραφο το οποίο παρουσίασε η Oxfam και τους συγχαίρω για την εργασία τους. Και τέλος θέλω να πω ότι βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον από τα τρία θεσμικά όργανα αλλά δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε δράση, χρειαζόμαστε ε, χρηματική βοήθεια και επιπρόσθετη συνδρομή και γι' αυτό κυρία Πρόεδρε τώρα θα ακούσω. Θα συναντηθώ την Τετάρτη με τους σκιώδεις εισηγητές και την Πέμπτη το απόγευμα είμαι ε, ελεύθερος για όποια ε, μη κυβερνητική οργάνωση θέλει να με συναντήσει και να μου κάνει κάποια παρουσίαση. Ευχαριστώ. Και το λόγο έχει τώρα η κυρία Φρονσουάς Μωρό για πέντε λεπτά. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω να κάνω σε πέντε λεπτά είναι να σα εξηγήσω όλη τη διαδικασία προπαρασκευή στην Κομισιόν προκειμένου να γίνει αυτή η αναθεώρηση του 2010 των στόχων της χιλιετίας. Έχουμε το πακέτο επικοινωνίας το ΕΑΡΙΝΟ, Απρίλιος-Μάιος. Και έχουμε μια γενική μέθοδο εδώ. Το πακέτο αυτό είναι μια μεγάλη παλέτα θεμάτων βελτίωση της πολιτικής μας σε ορισμένους τομείς κλειδιά υγεία, εκπαίδευση, επιστημιστική ασφάλεια. Σύντομα θα έχετε έγγραφα και ανακοινώσεις για τα θέματα αυτά. Μελετάμε την επίπτωση των πολιτικών μας στην, στο να, είναι, να υπάρχει ακολουθία στις διάφορες πολιτικές. Εδώ και μερικές εβδομάδες εκπονούμε ένα πρόγραμμα εργασίας όπου σε σχέση με το γενικό πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν θα εντοπίζει τις πρωτοβουλίες που θα έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα θα είναι εργαλείο έγκυρης προειδοποίησης για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε σχέση με τις διάφορες επιμέρους πρωτοβουλίες. Τρίτο σκέλος της προπαρασκευής είναι η χρηματοδότηση. Τι κονδύλια χρειάζονται. Καταρχήν πρέπει να, δούμε, να το συγκρίνουμε με τους στόχους που έχουμε, την κλασική ετήσια έκθεση Monterey, κατά πόσον τηρήθηκε η διαδρομή, η κίνηση σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια. Δεύτερον, η δημοσιονομική χρηστή διακυβέρνηση και πόσον σωστά χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι για την καταπολέμηση των παράνομων ροών. Το συζητήσουμε στην άτυπη συνάντηση υπουργών στην Κράνχα, όπου κυρία Πρόεδρε είχατε την ευκαιρία να συμμετάσχετε. Και τρίτο σκέλος, οι καινοτόμε πηγές. Δηλαδή, τι δυνατότητες υπάρχουν στα πλώσια των διαφόρων τεχνικών ομάδων διεθνώς που ασχολούνται με το θέμα αυτό να αξιολογηθεί το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο το α ή το β μέτρο για κινητοποίηση επιπλέον πόρων. Ένα τμήμα των ανακοινώσεων θα τα έχουμε ήδη το Μάρτιο. Το υπόλοιπο πακέτο <clears throat> θα εγκριθεί και θα σταλεί από την Κομισιόν στις 21 Απριλίου και μετά. Στόχος όλων αυτών των μέτρων είναι θέση της Ένωσης με πλήρη ακολουθία σε σχέση με όλα τα σημαντικά διεθνή γεγονότα αποφασιστικά για τη λήψη των αποφάσεων όπως η διάσκεψη Ένωση Αφρική τέλος του χρόνου πιο πριν η διάσκεψη των G8, των G20 έτσι ώστε να υπάρχει μία θέση της Ένωσης με πλήρη συμφωνία με όλα τα άλλα επιμέρους στοιχεία και όσο πιο φιλόδοξη γίνεται. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Η κυρία Νίκολα Χάρινγκτον. Πέντε λεπτά παρακαλώ. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ευκαιρία γιατί υπήρξε και για προτεραιότητα του Γενικού Γραμματέα, όχι μόνο το 2010, αλλά και για όλη αυτή την περίοδο μέχρι το 2015. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τους στόχους του κυρίου Γενικού σε συνάντηση υψηλού επέδου, τη διαδικασία της προπαρασκευής και αυτό το οποίο ζητεί από τις αντισόμενες ε, αναπτυγμένες ε, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Ε, UNICEF, ILO, ε, UFPA, όλες αυτές οι, όλοι αυτοί οι φορείς ε, ε, ανταποκρίνονται και νομίζω ότι όλοι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή την έκθεση. συμφωνούμε επομένω ότι η διακήρυξη αυτή των στόχων της χιλιετίας είναι μια δέσμευσή μας, δικαιώματα, ανάπτυξη και θα πρέπει πρέπει να παίξει το ρόλο της η η Ευρώπη και δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύη, είναι και δικό τη συμφέρον. Είναι σαφές το μήνυμα. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε τον του 2015. Θα πρέπει να μην αναβάλουμε και να κάνουμε αυτό που πρέπει σήμερα σε σχέση με τις υποσχέσεις μας. Οικονομική κρίση, αλλαγή κλίματος, διατροφική κρίση, όλα αυτά μπορούμε να πατύχουμε αυτούς τους στόχους μας ε, θα χρειαστεί παραπάνω προσπάθεια και στοχευμένη δράση. Επίση, έχουμε αυτή την συνάντηση του επίπεδου που νομίζουμε ότι είναι μοναδική ευκαιρία τόσο να μπορέσουμε να ενισχύσουμε προσπαθίε μα και να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση στο στόχο του 2015 να βρούμε πού υπάρχουν κενά, να μπορούμε να, ε, να δούμε ποιε είναι προτεραιότητε, να μπορέσουμε επίση να αναλάβουμε δράση. Επίση, μα λέει συγκεκριμένα ο κ. Γενικό ότι θα πρέπει να έχουμε μια ατζέντα δράση 2015-2015 μέχρι το 2015 τέλο πάντων, ούτω ώστε να μπορέσουμε να δούμε ε, τι χρονικά πλαίσια θα έχουμε, τι, τι, θα, τι μηχανισμούς θα βρούμε, ούτω ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ο ΙΕ, να βοηθήσει και την Ευρώπη, αυτούς που βλέπουν τις και το Κοινοβούλιο. Και έχουμε και αυτή την ε, έκθεση του κύριου Γενικού του Τελημαρτίου που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε ε, τι πήγε καλά και τι δεν πήγε καλά. Διότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι ε, να δούμε κάποια συμπεράσματα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε κάποιες συστάσεις, να είναι πιο καλή η συνεργασία. Και η Διευθύνουσα Ομάδα για την Αφρική επίσης θα μας δώσει κάποιες ιδέες γιατί ξέρουμε ότι ε, θα μπορούσαμε να βρούμε εκεί πέρα τι προβλήματα έχουν σε σχέση με τους στόχους αυτούς. Έχουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει για την προπαρασκευή ε, της συνάντησης αυτής και έτσι έχουμε και την ε, ε, ατζέντα δράσης του κυριογενικού ούτω ώστε να μπορέσουμε δυναμικά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και θεωρούμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια βασικά σημεία για διερεύνηση, για διαβούλευση με το Κοινοβούλιο επίσης θέλουμε να έχουμε εκθέσεις ανά χώρα, ούτως ώστε να δούμε ε, τι θέλει κάθε χώρα, τι την προβληματίζει, τι τη ζητά και επίσης να μπορέσουμε να ελοπίσουμε τους ε, δείκτες, τους παράγοντες επιτυχίας. Τέλος, θα έχουμε κάποιες αξιολογήσεις τον Ιούνιο σε επίπεδο ε, του ΟΗΕ για τις υποσχέσεις της δεσμεύσης του Γκλενίγκλς. Ακόμα λοιπόν και στις χώρες που είναι ουραγοί τώρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα, ότι χρειάζονται παρεμβάσει, ούτω ώστε να γίνει κάτι για του στόχου τη χιλιετία. Τρει προκλήσει. Ε, εθνικά ε, πλάνα, χρηματοδότηση, αλλά και εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών της υλοποίησης. Επομένως, το βασικό είναι το πώς θα μπορέσουμε να μην χάσουμε το τρένο των αλλαγών τις επόμενες, ε, τα επόμενα χρόνια. Και χρειάζεται επομένω μια παρέμβαση, χρειάζεται μακρόπνοη δράση, στρατηγικές και έτσι να έχουμε βιωσιμότητα. Και αυτές οι επιταχυνόμενες δράσεις σημαίνει ότι θα πρέπει να βοηθήσει η γεωργία, ε, ε, παιδεία, υγεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το θέμα στις ε, διαστάσεις. Και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε αυτό το οποίο θέλουμε με συνεργασίες. Και στην εκθεσή του ο Γενικός θα πει ότι υπάρχει παγκόσμια κρίση. Και με ορίζοντα 2015 θα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας για την ενίσχυση, την αρρωγή, την άρση των χρεών τον ε, Ιούλιο, πέρσι αλλά και φέτος έχουμε αυτά τα κείμενα τα οποία ξεκαθαρίζουν το τι οφείλουμε να κάνουμε. Άλλα τέσσερα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να τα κάνουμε για να είναι επιτύχει των στόχων. Οι στόχοι θα περισσότερο λόγω της κρίσης. Όμως, σε σχέση με άλλους στόχους θα είναι πιο μικρή η δαπάνη. Για ομονές χώρες θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των, περιστάσεων και να προσέξουν το θέμα των επιδοτήσεων και τη σβήσιμο της ε, φτώχειας. Όλα αυτά ε, είναι προβλήματα σε πολλές χώρες. Και λόγω αυτής της κρίσης χρειάζεται χρηματοδότηση, πάγωμα χρεών, πάγωμα και αναδιάρθρωση του χρέους για τις χώρες που έχουν πρόβλημα. Η τεχνολογία να την εκμεταλλευτούμε για να σβήσουμε τη φτώχεια. Τι άλλο μπορεί να κάνει η Ευρώπη. Εν κατακλείδη κυρία Πρόεδρε, να σας φέρω τα να μπορέσει να τηρήσει τις υποσχέσεις να κάνει αυτά που λέει ο ΙΕ για αυτή την ανάληψη δράσης. Αφετηρία θα είναι οι σημερινές υποσχέσεις και να δουν οι άλλες χώρες ότι τηρεί τις υποσχέσεις της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό. Και έτσι να ε, υπάρχει κάποια ενεργή συμμετοχή σε αυτή την συνάντηση υψηλού επίπεδου και έτσι να έχουμε κάποιες διακρατικές συμμαχίες για την υλοποίηση αυτής της ατζέντα προοδευτική είναι αυτή η πολιτική που να μας βοηθήσει να πετύχουμε τους αναπτυσιακούς αυτούς στόχους της χιλιετίας. Μία τελευταία σκέψη, Πρόεδρε. Αυτή η συνάντηση θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, αλλά υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Είναι θέμα αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών. Γιατί χρειάζονται την ανάπτυξη για αναπτυγμένες χώρες, για αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά είναι και θέμα της αξιοπιστίας ε, των ανεπτυγμένων χωρών και του ίδιου του ΟΗΕ που χρειάζεται την στήριξή σας. Ευχαριστούμε. Έπρεπε να σας κόψω, να σας σταματήσω, να σας αφαιρέσω το μικρόφωνο γιατί πέρασατε κατά πολύ το όριο των τριών λεπτών. Oxfam. Έχετε 7 λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στην Oxfam International θεωρήσαμε την πάρα πολύ σωστή ευκαιρία μας δώσατε σήμερα να σας μιλήσουμε και εμείς, όπως και εσείς, έχουμε κοινούς στόχους, ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολέμηση φτώχειας το 2010. Πάρα πολύ κρίσιμη χρονιά. Και αυτό η έκθεση Κάσμαν θα είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για την ανάλυση δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις γιγαντιές προκλήσεις. Πέρσι ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Σε βορρά και νότο. Δυστυχώς ο καθένας έχει άλλη αντιμετώπιση στα προβλήματα αυτά. Οι πλούσιοι βρήκαν κάποια αποτελεσματικά μέτρα για κοινωνική πρόνοια και οικονομική σταθερότητα στις χώρες τους. Όμως, ο ΙΕ, το G20, οι άλλοι φορείς δεν κάνανε πολλά πράγματα για τις συνέπειες αυτής της κρίσης σε φτωχές χώρες. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι χρειάζεται κάτι να γίνει. Έχουμε αυτό το 1,4 δισεκατομμύρια που ζουν σε βαθιά φτώχεια. Το τώρα λέει ότι 90% των Ευρωπαίων είναι υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας. Άρα, θα πρέπει όμως αυτό να είναι κάτι που θα το προβάλλουμε, να είναι ορατό. Όλοι επομένω έχουμε στρατευτεί. Να ακουστεί η φωνή μας και να είναι ενιαία, με μια φωνή να μιλήσουμε. Έχει πάρα πολύ καλή το ότι θα κάνετε εσείς για να πειραστεί οι, οι κυβερνήσεις. η διακήρυξη για τους στόχους της χιλιετής είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε θα χάσουμε αξιοπιστία σχέση με τους ε, στόχους που ήδη ετάξαμε και, και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι θα έχουμε αποτύχει. Αλλά αποκλείεται να αποτύχουμε. Δεν Αυτό το σενάριο αποκλείεται εν ώψη του Σεπτεμβρίου. Πολύ μεγάλη ευθύνη. γιατί έχουμε η ίδια τάξη κάποιες ευθύνες που φέρουμε και δεσμεύσεις. Για πρώτη φορά οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας θα πάνε σε αυτές τη συνάντηση με κοινή θέση. Πώς θα πετύχουμε όλοι τους στόχους. Η ΕΠΑ επίσης κινούνται στην κατεύθυνση. Και η Ευρώπη ήδη έχει επενδύσει σε αυτό να τιμήσουμε αυτές μας τις συνδέσεις, να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα, τι χρειάζονται αυτοί οι 1,4 δις άνθρωποι που ζουν στη φτώχεια. Δεν χρειάζονται δηλώσεις καλής θέλησης. Ούτε ανακύκλωση. Θέλουν συγκεκριμένες πράξεις, δράσεις, άμεσης υλοποίησης με συγκεκριμένα κριτήρια. επίτευξη ενός ή δυο τομιακών στόχων δεν αρκούν, γιατί δεν ζει με τομιακές επιτυχίες ο κόσμος. Χρειάζεται ένα σφαιρικό σχέδιο με εγκάρσιους στόχους. Άρα, το θέμα δεν είναι περισσότερα χρήματα. Το θέμα είναι πώς θα είναι πιο ποιοτική προσπαθία μας. Συνεπής πολιτική, αποτελεσματική πολιτική, αξιοποίηση των ιδίων πόρων αυτών των χωρών του Νότου. Οι φτωχοί δεν χρειάζονται διανομενίστικα λόγια για το τι πάνε τι εγγύησε, τι θα γίνει το 2015. Χρειάζονται αποτελέσματα εδώ και τώρα. Και αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό είναι οι προτάσεις μας στην Oxfam. Έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε προς την επίτευξη των στόχων τη χιλιετία και να είναι τα βήματα μας σαφή και ξεκάθαρα πρώτα-πρώτα να βελτιώσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή για την επίτευξη των στόχων. Για πιο συγκεκριμένα ε, έχουμε τα εξή τρία σημεία. Δημοσιονομική στήριξη, 50% της ενίσχυσης για συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2015 αργότερο. Δεύτερον, αν μελη θα πρέπει να εισφέρουν μέχρι το 15% ε, των ε, εισφορών τους ή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Τρίτον, κατανομή της εργασίας του έργου σημαίνει ότι θα πρέπει κάποιους παραμιλημένους στόχους να τους ξαναενεργοποιήσουμε ας πούμε τα της υγιεινής προς μέρες μητέρες, ανήλικους και άρα να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες συμφωνίες εταιρικής σχέσης για την προαγωγή αυτών των στόχων. Επίσης, πολυμερή μέσα χρηματοδότησης. Συντονισμός με τις χώρες αυτές. Όπως η ταχεία πρωτοβουλία για την παιδεία. Ή επίσης αυτά τα κάθετα κονδύλια για την υγεία. Τα στοιχεία του 2010, οι στόχοι, οι ποσοτικοί μάλλον δεν θα καλυφθούν, αλλά είναι θέμα αξιοπιστής Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι επιγόντως χρειάζεται νομοθεσία δεσμευτική, εθνική νομοθεσία ούτως ώστε να μπορέσουμε να τιμήσουμε αυτές μας τις δεσμεύσεις για τη χιλιετία. Τέταρτον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι επιπλέον χρηματοδότηση όπως προανέφερα. Το 0,7 δεν φτάνει. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει περισσότερα χρήματα από όλες τις κατευθύνσεις. Ειδικού φόρους. Και πάγωμα του χρέους για αυτές τις χώρες που χτύπησε πιο σκληρά η κρίση. Έτσι θα πιστεύουν τους στόχους της χιλιετίας. Μας λένε ιδεαλιστές, εθροβάμονες, ουτοπιστές. Τα ίδια λέγανε όμως και για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο των Εγκλημάτων Πολέμου. Να, όμως που τώρα κάποια όνειρα έχουν υλοποιηθεί. Αποφασιστικότητα έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβουλίο σας. Γι' αυτό και ευθυνόμαστε σε εσά. Δείξτε την ίδια αποφασιστικότητα. Έχουμε αυτή την πρόκληση για το 2010. Θυμάστε εκείνη την άσπρη κορδέλα γύρω-γύρω από το κοινό του 2005, ούτως ώστε να δηλώσουμε, να διακηρύξουμε ότι καταπολύουμε τη φτώχεια. Το ίδιο πρέπει να γίνει και τώρα. Μεγάλη πρόκληση, μεγάλες προσπάθειες που απαιτούνται. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Και τώρα οι συνάδελφοι έχουν το λόγο. Ο κύριο Γκέρνη πρώτο. Ευχαριστώ. Θα περιοριστώ στα οικονομικά. Όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων τη χιλιετία. Ακούσαμε την εκπρόσωπο τη Oxfam. Συμφωνώ εν πολλής με την άποψη αυτή. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές. Ποιος έχει την ευθύνη αν υπάρξει αποτυχία. Γιατί οι στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη δεν αφορούν μόνο την Ένωση. Η Ένωση είναι ο κύριος χρηματοδότης. Το θέμα είναι ποιος θα κάνει τι και τι συμφωνεί με τις υποσχέσεις που δόθηκαν το έτος 2000. Ας πούμε ότι η Ένωση δεν θα είναι στο ύψος των υποχρεώσεων της, των δεσμεύσεων της, αν δεν δώσει τα ποσά που έχει υποσχεθεί. Πρώτο γενικό σχόλιο. Μία ερώτηση από αυτού. Στο βαθμό που η Ένωση συμμορφωθεί με τις οικονομικές δεσμεύσεις της που επαναλήφθηκαν και στην Ευρωπαϊκή Ομοφωνία όσον αφορά την ανάπτυξη δεν θα είναι στο ύψος της υποχρέωσής της όσον αφορά το σύστημα νέου χαρακτηρισμού της βοήθειας. Δηλαδή στην Κοπενχάγη μερικές κυβερνήσεις παρέμειναν ασαφείς ως προς το ότι τα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια συμφωνούν με τους στόχους της ανάπτυξης της χιλιετίας και θα πρέπει να παραμείνουν προς το στόχο αυτό ή θα έπρεπε να δοθεί μια νέα ετικέτα σε σχέση με το χρέος το οποίο συνήψε η Ένωση προκειμένου να μετριάσει την επίπτωση της οικονομικής κρίσης και της αλλαγής του κλίματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εγώ δεν θέλω να παίρνω μέρος σε μια μέθοδο αυτομαστίγωσης. Από τη στιγμή που έχει αναλάβει μια δέσμευση κομισιόν πρέπει και εμείς να συστοιχηθούμε με την ε, Κομισιόν και να υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα, ποσοστά όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις. Και να πούμε ποιες χώρες μέλη είναι αυτές. Να πούμε ρητά ποιες χώρες συμμορφώθηκαν με αυτό που υποσχέθηκαν στην, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομοφωνίας. Σας θυμίζω ότι για το 2010 ο μέσος όρος είναι 0,56% του ΑΕΠ της Ένωσης και το 2015 0,7%. Συμμορφώνονται με αυτό ποιες χώρες μέλη και η Ένωση. Και να δούμε ποιες δεν συμμορφώνονται. Έχουμε μετά τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους που έδωσαν υποσχέσεις. Αυτά. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς. Ο κύριος Ντέβα. Ευχαριστώ. Μερικές ερωτήσεις. Συνεργαζόμαστε με το Ηνωμένα Έθνη, με τον Jeffrey Sachs, Quick Wings, έχουμε clusters, έχουμε ένα σωρό συστήματα. Μπορεί κάποιος να αναλύσει και να μας πει γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρξαμε επιτυχής και γιατί Υποθέτουμε ότι με διαρκή επιτάχυνση θα πετύχουμε σε πέντε χρόνια κάτι που δεν μπορέσαμε να πετύχουμε σε δέκα χρόνια. Θέλω μια λογική, πρακτική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όμως και τον Μάικλ Κάσμαν γιατί Ε, όπως και η εκπρόσωπη τη και το ΟΗΕ μας έκανε πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Ε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για, το 2010 αυτό το έργο που είχε αναλάβει η Επιτροπή μας. Το 2010 όπως είπε και ο Μάικλ ο κείμενό του το οποίο μας διαβίβασε, εμείς θα πρέπει να κάνουμε κάτι ως ανεπτυγμένες χώρες για κάτι που το υποσχεθήκαμε και είναι μια υπόσχεση μια συμβιβασμό, έχουμε κάτι συγκεκριμένο, συγκεκριμένη ρότα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το 2000 είπαμε ότι θα πρέπει να πάρει αυτή την κατεύθυνση ο ΙΕ και ε, μετά μέχρι το 2007 προχωρήσαμε αρκετά γρήγορα αλλά δεν άρκεσε αυτό. Οπότε ε, εδώ και, κάνα δύο χρόνια ε, εν ώψη των μελουσών εξελίξεων έχουμε το πρόβλημα του ότι μπορεί να ε, επιβραδυνθούμε, μπορούμε τελικά να βρεθούμε μακριά από την επίτευξη των στόχων που έχουμε εντάξει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η Ευρώπη θα πρέπει να είναι η ατμομηχανή, θα πρέπει να είναι ο θετικός καταλήτης για αυτό που προσπαθεί να κάνει ο ΙΕ. Μόλις σήμερα εγκρίναμε στην Επιτροπή μας αυτό το κείμενο που αφορά την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων όσον αφορά την θέση, την τοποθέτηση ε, που θα λάβει εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνοντας υπόψη κάποια, θέματα που έχουν να κάνουν με τους στόχους της χιλιετίας. Ε, τώρα προσπαθούμε να εκπονήσουμε κάποιες πολύ σημαντικές εκθέσεις στην Επιτροπή μας Φερρυπίν η έκθεση της Φραντσέσκα Κέλλερ όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και συνέπεια της ε, αρρωγής. Πολύ σημαντικές υποθέσεις, ούτω ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε τους στόχους που θέλουμε. Όμως, επίκεντρο όλων αυτών θα είναι η έκθεση Κάσμαν και για την Επιτροπή μας και για το Κοινοβούλιο, ούτως ώστε έτσι να διαμορφωθεί μια θέση πριν την Ιαρινή Σύνοδο του Συμβουλίου. Επίσης, ξέρω ότι ενδιαφέρεται η Ισπανική Προεδρία θα πω ότι θέλει το Ιερινό Συμβούλιο να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς την συνέλευση του ΟΗΕ. Θα βοηθήσω όσο μπορώ τον Μάικλ. Και έτσι η έκθεσή του να αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη θέση της Ευρώπης, ούτω ώστε να προχωρήσουμε σε μια επαναδιατύπωση των στόχων της χιλιετίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα συμπληρώσω τον κύριο Κάσμαν στη σχέδιο έκθεσής του και τους έντονους τόνους που χρησιμοποιεί. Σχεδόν μη κοινοβουλευτική είναι η όρη αυτή. Μου αρέσουν όμως. Ήρθε η ώρα για δράση. Αναφέρεται σε, σε άλλα θέματα κλειδιά πολιτική ανάπτυξης. Θα ήθελα να είμαστε σαφείς στην Επιτροπή μας. Ότι για να πετύχουμε πρέπει να υπάρχει ακολουθία στη δράση μας. Φερρυπίν, στην Αλία το Κοινοβούλιο ψήφισε ότι η αλληλευτική μας πολιτική καταρχήν θα πρέπει να ωφελεί τους αλλιείς στην Ευρώπη. Κατ' εμέ είναι κατά τη συνθήκη της Λισαβόνας, άρθρο 2.8, που λέει ότι οτιδήποτε στην εξωτερική μας πολιτική δεν πρέπει να παραβλάπει την ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν υπάρχει στη συνθήκη της Λισαβόνας. Και συμφωνώ με τον κύριο Κάσμαν ότι πρέπει να το πούμε αυτό. Και έχω και μία ερώτηση και προς τον εισηγητή και στους, ε, στους που μίλησαν μέρους της Oxfam για την δημοσιονομική υποστήριξη. Ναι, να έχουμε υποστήριξη 50% του προϋπολογισμού. Η υποστήριξη του προϋπολογισμού είναι χρήσιμη, αλλά σημασία έχει ο ορισμός. Εγώ είμαι Ολλανδέζα και ξέρω ότι η κυβέρνησή μου είναι υπέρ της δημοσιονομικής υποστήριξης, αλλά όχι όπως το κάνει η Κομισιόν. Γιατί αυτό γίνεται χωρίς κανόνες. Μπορεί να είναι λίγο έντονη αυτή η διατύπωση. Ωστόσο, ποιε χώρε, ποιοι κανόνε και γιατί ειδικά το 50%. Συνήθω η δημοσιονομική υποστήριξη είναι φτηνή για τη δίκηση της χώρα που τη δίνει τα χρήματα αυτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και αποτελεσματική στη χρήση τη. Θα ήθελα μερικά σχόλια και από τον Κάσμαν και από την Oxfam και την Intermont. Πρόεδρος. Ο κύριος Γκέρενς θέλει να προσθέσει κάτι. Ξέχασα μία ερώτηση προς την Κομισιόν. Επειδή στην Κομισιόν μοιράζεται το έργο σας, την Ευρωπαϊκή Χρηστή Διακυβέρνηση, θα ήθελα να ξέρω ποιος επίτροπος είναι ο κύριος υπεύθυνο για το συντονισμό όλων αυτών των μέτρων. Πρόεδρος. Άλλοι συνάδελφοι. Κανείς. Προς απάντηση των ερωτημάτων των βουλευτών ξαναδίνω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Η κυρία Φρασάς Μωρό. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για να απαντήσω στα ερωτήματα. Σας μίλησα για το πακέτο που ετοιμάζουμε υπό τον Επίτροπο Πίμπαλτς που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη και για τη σχέση με τις χώρες ΑΚΕ. Η κυρία Νίκολα Χάρινγκτον, δύο λεπτά. Δεν θέλει να... Η κυρία Χάρινγκτον, δύο λεπτά. Ευχαριστώ για να απαντήσω στο ερώτημα του Αντιπροέδρου. Υπάρχουν, έχει γίνει συλλογή στοιχείων για συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα μέρη. Και το θέμα είναι πώς θα διδαχθούμε από το τι θα χρειαστεί για να μεγεθυνθούμε, να έχουμε αντίδραση. Θα πάρουμε, αν θέλετε διμερώς αν θέλετε να συζητήσουμε τις περιπτώσεις αυτές όπου μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι σημειώθηκε πρόοδος. Μπορούμε να το κάνουμε διμερώς. Πρόεδρος, η κυρία Ιρέν Μιλέρο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να μιλάμε για αποτυχία αυτή τη στιγμή. γιατί, δεν να κάνουμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε σε πέντε χρόνια γιατί δεν μπορέσουμε να κάνουμε σε 10 χρόνια. Πρώτον, έχουμε περισσότερη εμπειρία. Δεύτερον, όταν τα πράγματα μα πιέζουν, δρούμε καλύτερα. Αν δούμε τι έγινε με τη διάσωση του οικονομικού συστήματος, βλέπω ότι όταν υπάρχει πολιτική βοήθεια για κάτι, γίνεται. Πρέπει να σεβόμαστε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, που δεν το κάνουμε στο παρελθόν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και να ασκήσουμε πίεση για υποστήριξη μέσω του προπολογισμού. Όντω υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό. Και αν θέλετε μπορούμε να σα στείλουμε περιπτώσεις. Είναι ένα από τα εργαλεία. Ένα εργαλείο προκειμένου να αποδοτικά να χρησιμοποιείται η βοήθεια από τη συγκεκριμένη χώρα και να αυξηθεί και το κυβερνητικό δυναμικό για την εκτέλεση. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα πώς λειτουργεί η υποστήριξη, σύστημα υποστήριξης του προϋπολογισμού. Το 50% ε, κάθε ποσοστό έχει ένα, μια διάσταση προσέγγισης. Λέμε 50% υποστήριξη του προπολογισμού θα ήταν καλό. Φαίνεται σαν να μιλάμε για MTGs από την σκοπιά του Βόρειου Μεσφαρίου. Ε, Περί το Μαρτίου ο κύριος Κάσμαν οργανώνει μια εκδήλωση εδώ στο Κοινοβούλιο όπου 8 γυναίκες θα από χώρες του Νότου και θα μας μιλήσουν για την επίπτωση της κρίσης στις χώρες τους και πώς μπορούν να βγουν από την κρίση αυτή και θα πάω να ακούσω, να δω τι έχουν να πούνε οι άνθρωποι από το Νότο και τι ζητάνε από την Ένωση να κάνει. Πρόεδρος. Κύριε Κάσμαν, έχετε το λόγο μερικά λεπτά για να κλείσουμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν σήμερα για τις ιδέες που εξέθεσαν. Όλοι κινούμαστε στον ίδιο δρόμο. Είπα προς την Κομισιόν και άλλους ότι όλες οι πολιτικές μας έχουν επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως ενέργεια, γεωργία, περιβάλλον, υγεία, μετανάστευση, αλληλεία και φυσικά οι εξωτερικές υποθέσεις. Όλες αυτές οι πολιτικές έχουν επίπτωση στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάγκη εκρίζωσης μια για πάντα της στέρησης και της φτώχειας, της ένδυας και της φτώχειας. Η έκθεση αυτή δεν είναι δική μου. Μετά από σειρά συναντήσεων τη συνέταξε ο κύριος Μόρμο, κάθε αριστερά σας κυρία Πρόεδρε. Η γραμματεία δηλαδή βόηθησε αφάνταστα και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Διαφορετικά θα είμαστε απλώς μαριονέτες Πρόκειται για ένα συνδυασμό δράσης. Γραμματεία, βουλευτές. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας μιλήσουμε για τις επιδοτήσεις που δίνουμε στην υπερπαραγωγή που πάει στις αναπτυσσόμενες χώρες και τους πίσω γυρίζει προς τη φτώχεια. Να δούμε τις αλλιαστικές συμφωνίες. Δεν έχει σημασία ποια χώρα μέλος. Όλα αυτά μετράνε. Και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει όημα να λέει ναι να συνεχιστεί η μη ηθική κοινή γεωρική πολιτική και από την άλλη μεριά να λέει ναι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης της χιλιετίας. Ευχαριστώ την κυρία Χάρινγκτον για τη δέσμευσή της και για το ότι μας εξέθεσε για τα προγράμματα, τα σχέδια μάλλον του Γενικού Γραμματέα ιδιαίτερα στην την εφαρμογή μια ανεπαρκής χρηματοδότηση επιτάχυνση της υλοποίησης και για τον αγαπητό μου φίλο Ντέβα που θέτει πάντα τις δύσκολες ερωτήσεις αλλά στο τέλος τελικά είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί για να πετύχουμε τους ίδιους στόχους. Ναι, οι δεσμεύσει πρέπει να τηρηθούν και συμφωνώ με τον κύριο Γκέρανς αλλά πρέπει να πάμε πιο πέρα από το 0,7% του ΑΕΠ και ταυτόχρονα να στυλιτεύσουμε αυτούς που δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν. βοήθεια ως προς το εμπόριο. Έχουμε το στόχο του 2015 και η Ευρώπη, η Ένωση, ως ο πιο μεγάλος χρηματοδότης του προγράμματος αυτού, καλείται να δράσει. Ευχαριστώ την όξφα μου, όπως είπα και πριν, για τη συμβολή σας, για το κείμενό σας. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Για τον κύριο Γκέρενς, έχει δίκιο. Τι κάνει ο Καναδάς, η Αμερική και οι άλλοι. Ας δώσουμε εμείς όμως πρώτοι το παράδειγμα. Και με το παράδειγμα αυτό ας στυλιτεύσουμε τους άλλους. Ας αποφανθεί η ιστορία. Ας κάνουμε εμεί τις αλλαγές που βελτιώνουν ζωές. Διότι κυρία Πρόεδρε, είναι ένα μωρό που κλαίει στην Αφρική έχει διαφορά με ένα μωρό που κλαίει στις Βρυξέλλες το παιδί ή το μωρό στις Βρυξέλλες θα μπορούσε να ήταν στην Αφρική θα μπορούσε να είναι το μωρό ή το παιδί στην Ασία ή στη Λατινική Αμερική ή στο Μπέρμιχαμ είναι η καθολικότητα αυτού που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο μπορεί εύκολα να συμβεί σε κάποιον άλλον που είναι λιγότερο ευνοημένος από τη ζωή. Ενρίκη, σε εναν ανθρωπο μπορει ευκολα να συμβει σε καποιον αλλον που ειναι λιγοτερο ευνοημενος απο τη ζωη ενρικη ευχαριστω για τη βοήθειά σου την δέσμευση να με βοηθήσει στην Ισπανική Προεδρία και είμαι σίγουρος ότι η Ισπανική Προεδρία θέλει αυτό να είναι επιτυχία. Αλλά έχουμε μερικές διστακτικές χώρες που ήδη λένε μας παίρνει οικονομικά να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε σε καιρούς κρίσης και όταν έχουμε το πρόβλημα με το κλίμα. Μα η οικονομική κρίση μας δίνει την ευκαιρία να ξαναρχίσουμε να ξαναδούμε τις καινοτομίε για τη χρηματοδότηση, για έναν επιπλέον φόρο ενδεχομένω στο εμπόριο, στα εμβάσματα που γυρίζουν στις χώρες αυτές που είναι πολύ περισσότερα σε ύψος από τις δωρεές και τη βοήθεια που στέλνουμε. Αρκεί τα εμβάσματα αυτά να μην τα περικόπτουν ορισμένοι. Judith Σαργεντίνη, συνάδελφο Σαργεντίνη, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη. Για την υποστήριξη μέσω του προπολογισμού. Αν αυτό ήταν η απάντηση, θα την είχαμε εφαρμόσει εδώ και χρόνια. Δεν είναι η μόνη απάντηση. Ίσως μέσω της υποστήριξης του προπολογισμού μπορούμε να αποτρέψουμε σπατάλες, επικάλυψη και να δώσουμε τη δυνατότητα στις συγκεκριμένες χώρες για λύση γιατί η ενίσχυση, η ανάπτυξη και το εμπόριο, αν δεν έχει εξουσία μια χώρα, δεν πετυχαίνει τίποτα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Τελειώνω όπως άρχισα. Είναι μεγάλο προνόμιο για κάποιον να του δοθεί η δυνατότητα να συντάξει αυτή την έκθεση. Πρόεδρος, λυπάμαι για το ότι η χώρα μου δεν είναι στο ύψος των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει και θα πιέσουμε τους υπουργούς μας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους σας και περνάμε στο σημείο 5 πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 1934-2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και λοιπές χώρες υψηλού εισοδήματος. Γραπτές τροπολογίες δεν έχουμε για την έκθεση ΔΕΒΑ. Ο εισηγητής προτείνει μερικές προφορικές τροπολογίες σε σχέση με άλλες επιτροπές, ΑΦΕ και ΙΝΤΑ. Έχετε πάρει ήδη τις προτάσεις του εισηγητή μας. Αν δεν έχετε αντίρρηση στις προφορικές τροπολογίες, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Άρθρο 1 σημείο 3 αποσύρεται. Άρθρο 1 προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται άρθρο 1 σημείο 3 σε 3 γάμα προφορική τροπολογία 2 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1 σημείο 3 δέλτα προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τελική υποφορία. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα μάλιστα κύριος Δέβα κάτι δεν πήγε καλά κάτι φαίνεται δεν πήγε καλά λέει ο κύριος Δέβα εξισύσθεση προς το Συμβούλιο σχετικά με την 65η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έκθεση Γκερέρο. Παράγραφος Α. Τροπολογία 2 προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ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 Donc, um... Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος α, τελευταία παύλα 4, προφορική τροπολογία 3, υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ συγγνώμη η προφορική τροπολογία 4 πρώτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 5 καταπίπτει 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 που γίνεται η παράγραφος δέλτα α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ομόφωνα. Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης σε αναπτυσσόμενες χώρες έκθεση γκέτερα Κάσμανα. Θα μπορούσαμε να την ψηφίσουμε ένα μπλοκ. Αμπλοκ μέχρι την παράγραφο 5, την πρώτη σελίδα δηλαδή. Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Όλη την πρώτη σελίδα λοιπόν. Μάλλον μέχρι την παράγραφο 4 δηλαδή οι τροπολογίες 17, 18, 19, 20, 21, 22 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η προφορική τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Το 23 και 24. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρώτη συμβιβαστική. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύο. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Δεύτερη λοιπόν προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Καταπίπτει. 27 αποσύρεται. Καταπίπτει. Επίσης το 28, το, το 29 Ωραία, τώρα είμαι στο 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 και 31 καταπίπτουν. Η 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 39 χωριστά πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 καταπίπτει 42 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, προφορική τροπολογία 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, προφορική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 καταπίπτει 55 εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές ε, ε, απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εδώ θα πρέπει να ξαναμετρήσουμε ποιος είναι υπέρ της 62 non oui si qui sont contre oui très κατά προφανώς απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για να το ξανακάνουμε για το 64. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Έχει κολλήσει το ε, απορρίπτεται 10 υπέρ 11 κατά 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 αποσύρεται προφορική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 χωριστή ψηφοφορία πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το εκτιμώντας 9 ε, ναι, ή να τα κάνουμε όλα μαζί μέχρι το 12 από το 9 έως το 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά θα πάρουμε ομαδικά από το 16 ε, από το 16 μέχρι το 8. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το 1, 2, 3 μπορούμε να τα κάνουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Παράγραφος 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5. Ίντα. Να κάνουμε το 5 έως το 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά Περνάμε στην ΕΚΟΝ. Στη ΕΚΟΝ. Πρώτη παράγραφος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρία. Μπορούμε ίσως να κάνουμε μαζί μέχρι το 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ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 αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά μπορούμε να ψηφίσουμε 15 έως 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μετά είκοσι έως 22 Λοιπόν, ας κάνουμε μία γραμμή τη φορά. 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 22. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. στο 23. Το ΕΛΚ ζήτησε χωριστή ψηφοφορία. Το 23. Την παράγραφο 23 διαγράφοντας τη λέξη rights. Λοιπόν, θα ζητήσω από τη γραμματεία να διαβάσει και τις δύο προτάσεις. Λοιπόν, καταρχήν χωρίς τη λέξη rights και μετά με την, ε, μόνο τη λέξη rights χωρίς την ψηφοφορία. sexual and reproductive health rights, which is key to attaining the MDH, points out that a healthy, strong workforce is a precondition for economic development. Donc, un premier... Καταρχήν λοιπόν, σε πρώτο η χωριστή ψηφοφορία ψηφίζουμε χωρίς τη λέξη rights. Συμφωνούμε λοιπόν να κάνουμε χωριστή ψηφοφορία. Καταρχήν τι ψηφίζουμε δηλαδή. Πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ και μετά δεύτερο μέρος με τη λέξη right. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 26 σε συνδυασμό με τις τροπολογίες 70 και 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ 30 έως 35 όλα μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μπράβο. Non, on a plein de surprises tout le temps qui n'ont pas été vues. Alors maintenant, nous allons voter sur le budget 2011, section 3, commission ligne directrice pour le budget 2011. Προπολογισμός για τη χρήση του 2011, τμήμα 3. Δεύτερη παράγραφος, Προπολογία παριθμών 1. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, ποιοι απέχουν, εγκρίνεται. Τροπολογία Τρία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Προφορική στο 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα όσον αφορά την τροποποιηθήσα πρόταση ψηφίσματος, ποιο είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Νομίζω τελειώσαμε, λέει ο Πρόεδρος. Επομένως, Απαλλαγή. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη 6, 7 και 8. Έκθεση Μίτσελ. Χωρί τροπολογίε. Επομένω. Επομένω ψηφίζουμε το σώμα του κειμένου. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές και εγκρίνεται. Παρακάτω. Bon. Alors donc, ces deux derniers votes ne figurent έχουμε άλλε και ψηφορίε που δεν είναι στη μέρα ε, σε διάταξη και τώρα το ανακαλύπτω όπως και εσεί. Και ε, λέει η γραμματεία, συμφωνείτε να ψηφίσουμε σήμερα αυτά τα κείμενα. Απαλλαγή για το Fed έκθεση Μίτσελ. Δεν έχουμε τροπολογίε. Συμφωνείτε, ναι, πολύ ωραίο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Άρα εγκρίνεται. Δεύτερον, για τον Γενικό Προπολογισμό Τμήμα 3, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απαλλαγή. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά αποχές, εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ. Μισό λεπτό να δούμε τις ημερομηνίες για την επόμενη μας συνάντηση. Κύριε Γκέρντς, θέλετε το λόγο. Ναι, έχω μία ερώτηση σε σχέση με την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Τι, τι πάει να πει αυτό το οποίο ψήφισαμε, γιατί δεν είναι στα πλαίσια του προπολογισμού το ΦΕΔ. Από εδώ πέρα μου σφυράει ο γραμματέας δεν έχουμε δημοσιονομικέ αρμοδιότητες, αλλά μπορούμε να δώσουμε την απαλλαγή. Για την εκτέλεση του προπολογισμού, λέει ο κύριο Γκέρνς. Για την εκτέλεση του προπολογισμού τους. Ναι, ναι. Και αυτό που θέλω να μάθω είναι εμείς δίνουμε απαλλαγή στην ε, Κομισιόν εάν έχει απαλλαγή με τη σειρά από τα κράτη-μέλη. Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα διοικητικά του EDF. Επομένως, η Κομισιόν είναι αρμόδια για να κάνει την απαλλαγή. Η επόμενη συνάντηση μας είναι στις Βρυξέλλες, στις 16 ε, 3 με 6.30 και στις 17 το μηνός από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Τέλος για σήμερα. Γεια σας.